Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η παρουσίαση που θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ε, project τα οποία έχουν, ε, θα επιλεγούν για το 2011. Είναι στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 ε, νομίζω ότι έχουμε κοντά μας τον ε, κύριο Πακέ, ο οποίος μοιάζει να έχετε συνεδριάσει μας πιο πολύ από ότι τα πραγματικά μέλη. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω στην Επιτροπή σας και να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής ε, για την ε, ετήσια προκήρυξη για το Horizon 2020. Έχουμε ήδη παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πολιτούς προγράμματος για τις αρτηρίες της θάλασσας και για κάποια άλλα σημεία. Σας τα παρουσιάσαμε. Τώρα θα σας παρουσιάσω το ετήσιο και θα καλύψουμε, όπως θα σας περιγράψω, αρκετές προτεραιότητες από το χώρο των μεταφορών, αλλά θα εστιάσουμε και στο πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε το έργο αγωγή και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε περισσότερο αποδοτικοί για το Connecting Europe. Με συγχωρείτε που το έφερα μόλις τώρα, αλλά θα σας μοιράσω ένα φυλάδι με τα αποτελέσματα της επιλογής και δυστυχώς επειδή γίνεται σε πραγματικό χρόνο δεν μπορούσαμε να σας το στείλουμε πιο εμπρόθεσμα. Έχουμε πάντως συμπληρώσει κάποιες πληροφορίες στο φυλάδι, Αν ανατρέξετε στη σελίδα 39 θα δείτε πως γίνεται και μια λεπτομερής παρουσίαση των ε, project τα οποία εμείς ε, συστήνουμε για χρηματοδότηση. Έχετε λάβει όλο το έγγραφο αυτό, διακόπτει ο Πρόεδρος. αυτό είναι, πολύ ωραία. Όποιος δεν έχει παρακαλώ να ζητήσει από τη γραμματεία, είναι αυτό το οποίο σας δείχνω. Ωραία. Θα λάβετε κι εσείς το αντίτυπό σας. Συνεχίζει ο μελητής, συμπληρώσαμε με περισσότερες προφορίες από την περασμένη φορά, έτσι ώστε να έχετε αρκετές πληροφορίες για τα project προς χρηματοδότηση, αλλά προσπαθήσαμε να συμπληρώσουμε και μεγάλες πληροφορίες για τα έργα τα οποία δεν προτείνονται για χρηματοδότηση και μια σύντομη περίληψη της αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των πάνελ και για το πώς αποφάσισαν για το κατά πόσο θα προτείνουν ή όχι τη χρηματοδότηση. Κατά τη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την στήριξη της σχετικής εκτελεστικής υπηρεσίας και με τους εξωτερικούς αξιολογητές έκλεισε τη διαδικασία επιλογής και η απόφαση ε, που έχει 74 προτάσεις προς χρηματοδότηση, παρουσιάζονται στην Επιτροπή τους, θα παρουσιαστούν και στην Ολομέλεια, θα περάσουν ε, και την 5η 12 ε, Ιουλίου από την Financial Assistance Committee των κρατών μελών και μόλις λάβουμε την έγκρισή τους θα προχωρήσουμε με τη συνήθη διαδικασία διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τα τέλη του μήνα. Η απόφαση μετά θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση και η τελική απόφαση χρηματοδότηση για τα 74 αυτά έργα θα συζητηθεί με όσους τα προωθηθούν και για κάθε ένα ξεχωριστά θα λάβει ξεχωριστή μεμονωμένη απόφαση χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση πριν από τα τέλη της χρονιάς. Όπως σας είπα, για το 2012 είχαμε το πολιετές πρόγραμμα, τώρα έχουμε το ετήσιο μπροστά μας και η διάστρωση αυτού ε, επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τα όσα είχαμε στο περσινό ετήσιο Έχουμε πέντε βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η χρηματοδότηση για έργα τα οποία προωθούν την ολοκλήρωση των μεταφορικών συστημάτων. Είναι εκεί λοιπόν τα πολυμεσικά, είναι τα project για διασύνδεση, ε, η σύνδεση μεταξύ οδικών αξώνων και λιμένων για παράδειγμα. Η δεύτερη προτεραιότητα έχει να κάνει με την ελάφρυνση της ε, κλιματικής αλλαγής και με τα αέρια του θερμοκηπίου φαινός και καλύπτει επίσης και μια σειρά από έργα τα οποία προετοιμάστηκαν στα πλαίσια της συζήτηση που έγινε ε, για τις βόρειες θάλασσες, για τις ζώνες χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται αλλάζοντας τα καύσιμα για παράδειγμα ή με κάποια συστήματα επιστημονικά τα οποία θα επιτρέπουν να περιορίσουμε τα προβλήματα της ρήπανσης από θείο. Τουλάχιστον επαναλαμβάνω στις περιοχές όπου βρήκαμε ε, μεγάλη περιεκτικότητα. Είναι δηλαδή το υγροποιημένο αέριο, LNG και και όχι μόνο παρόμοια προϊόντα. Η τρίτη προτεραιότητα συζητήθηκε στα πλαίσια της, ε, του μέσου Connecting Europe για να βοηθήσουμε τους δικαιούχους να προετοιμάσουν τα έργα τα οποία καταθέτουν. Έτσι έχουμε λοιπόν το Project Pipeline το οποίο συνεχίζει να οριμάζει στα πλαίσια του Connecting Europe και έχουμε επίσης και μια σειρά αποστοχευμένα έργα όπου Χρειάζεται επίσης και, σκληρή, ε, ε, και σκληρές επενδύσεις στα πλαίσια του TEN-T. Όχι στα πλαίσια μόνο αυτού του μέσου, αλλά και στα πλαίσια των ομολόγων έργων, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε εμείς όσους έχουν σκοπό να βρουν καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω κάποιου πιο καινοτόμου μείγματο ιδιωτικών και δημοσίων κονδυλίων. Και εδώ ακούσαμε και κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις τέλος, αλλά όχι ίσονος σημασίας, γιατί πιστεύω ότι εδώ οι προτάσεις ήταν λιγότερε από αυτές που, είχαμε, που αναμέναμε. Το 5, η προτεραιότητα 5, ε, προετοιμάζει το έδαφος για το μελλοντικό TNT, που συζητήθηκε και εδώ στην Επιτροπή μας, συζητήθηκε και στο Συμβούλιο και προετοιμάζει το έδαφος κυρίως για την εφαρμογή των βασικών ε, αξώνων που αν επιβεβαιωθούν από ε, το Κοινοβούλιο θα αποτελέσουν και το βασικό μέσο και εργαλείο για να στηρίξει αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν θα χρηματοδοτηθούν δικαιούχοι οι οποίοι θα προετοιμάσουν το έδαφος για αυτούς τους διαδρόμους που είναι τόσο κομβικής σημασίας. Και βέβαια έχουμε εδώ πέρα και τους ε, άξονες τους, ε, που συνδέουν σιδηροδρομικά αυτά τα κομβικά σημεία, άρα λοιπόν θα υπάρχει και σιδηροδρομική διάσταση. Στο TNT έχουμε επικεντρωθεί σε κάποιες πολιτικές προτεραιότητες, αλλά προσφέρουμε παράλληλα και χρηματοδότηση για κάποια έργα ε, κατασκευαστικά. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. 200 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα. Προτάσεις και αιτήματα για χρηματοδότηση ύψους 426 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν υπερπλήρωση Είχαμε 100% αύξηση της έτσι, για χρηματοδότηση από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και αυτό είναι εξαιρετικό βέβαια γιατί έτσι εξασφαλίζουμε πως είναι τα καλύτερα έργα τα οποία προτείνονται για να χρηματοδοτηθούν. Όπως ε, συνήθως ακολουθήσαμε μια ε, διαδικασία σε δύο βήματα. Καταρχήν εξωτερική αξιολόγηση όπως ε, υιοθετήσαμε το πρόγραμμα το 2007 όπου εμπειρογνώμονε στον κλάδο των μεταφορών μαζί με την εκτελεστική υπηρεσία εξετάζουν τα έργα, τη συμμόρφωση αυτών με ποιοτικά κριτήρια, με την σχετικότητα με το TNT, με την προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την οριμότητα αυτών. Αυτή η εξωτερική αξιολόγηση μείωσε τον αριθμό των προτάσεων από τις 138 στις 84, δηλαδή 54 δεν προτάθηκαν για χρηματοδότηση από τους εξωτερικούς αξιολογητές γιατί δεν ανταποκρίνονται στα ε, κριτήρια κλειδιά από τότε που αποφασίσαμε να κάνουμε και την εξωτερική αξιολόγηση όπου σε βάθος αναλύονται ε, όλα τα, όλες οι προτάσεις έργου πρέπει να σας πω πως δεν έχουμε χρηματοδοτήσει καμία που να μην προτάθηκε από την εξωτερική αυτή τους εξωτερικούς αξιολογητές. Μετά, Περνάμε στη δεύτερη φάση, εξετάζουμε αυτές τις 84 προτάσεις για χρηματοδότηση. Πάλι είμαστε εκτός δυνατοτήτων προπολογισμού και εδώ έχουμε το εσωτερικό πάνελ με συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες, κομισιόν, Regio, Envy, Move, Γενική Διεύθυνση Move και με τη στήριξη της υπηρεσίας μας. Κοιτάξαμε τα έργα τα οποία είχαν προταθεί για χρηματοδότηση και προτείναμε 74 από τα 84 για χρηματοδότηση. Το οποίο σημαίνει ότι έχω, καλύπτουμε και τις πέντε προτεραιότητες της προκήρυξης. Σε κάποια τμήματα ήμασταν πιο επιτυχείς ε, από ό,τι σε άλλα. Τα στοιχεία αυτά σας τα δίνουμε στην πρώτη σελίδα του φυλαδίου και αν κοιτάξετε και τη σελίδα 10 θα διαπιστώσετε πως κατανέμει έτσι με εύκολα αναγνώσιμο οπτικό τρόπο τη γεωγραφική τοποθέτηση αυτών των έργων. Βλέπετε λοιπόν πως έχουμε μια καλή διάδοση στα κράτη-μέλη και αν δείτε και τα χρώματα θα δείτε σε ποια προτεραιότητα ανήκει το καθένα, το μέγεθος του ε, προπολογισμού που προτείνεται κτλ. Άρα λοιπόν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα είναι το μέσο έτοιμα και μετά η κατανομή επαναλαμβάνω πάει σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά. το 2012 θα, έχουμε, θα ανοίξουμε μια νέα προκήρυξη. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε άλλα έργα για το 2012, αλλά θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι μέχρι τα τέλη της χρονιάς και αν θέλετε θα έρθουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νέα προκήρυξη που θα είναι αυτή τη φορά πολυετής και θα χρησιμοποιήσει τον υπολείποντα προπολογισμό του προγράμματο και κάποιο τμήμα του προπολογισμού που θα απελευθερωθεί μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση για το πολιετέ και για το ετήσιο. Με συγχωρείτε για το πελιωτέ μόνο. Αλλά θα περιμένουμε κάποιο χρόνο ακόμα να ξέρουμε πόσο μεγάλη θα, αυτή, θα είναι αυτή η αναθεώρηση. Πάντως είτε φέτο είτε του χρόνου θα σα καταθέσουμε ένα τελευταίο πολιετέ πρόγραμμα, παρόμοιο με αυτό που σα παρουσιάζω σήμερα, όπου και πάλι θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στην προετοιμασία των project που είναι στα σκαριά και το πώς συνδυάζονται με τα TNT γιατί ελπίζουμε πως ε, θα είναι καλύτερη η συμμετοχή όλων των κρατών μελών, ευρύτερη, καλύτερη προετοιμασία έτσι ώστε τα έργα αυτά να συμπεριληφθούν τώρα, να ενταχθούν τώρα και να, όταν φτάσει η στιγμή να έχουν ε, οριμάσει όσο βρίσκονται στη διαδικασία ε, του pipeline, στα σκαριά δηλαδή. Ελπίζω λοιπόν πως για κάποια από αυτά μπορώ να τα μπορούμε να τα πούμε και μια επόμενη φορά, εάν θεωρείτε πως αυτό είναι ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κύριε Πακή. Θα τα δούμε λοιπόν ε, με τα μέλη. Κύριε Κάντιαν, για το ΕΛΚΑ. Δεν ξέρω αν εκπροσωπώ το ΕΛΚ, αλλά παρόλα αυτό θα πω όσα σκέφτομαι. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε ερωτήσει στον κύριο Πακέ. Βλέπω ότι μας παρουσίασε μια πολύ καλή δουλειά. Σε ό,τι αφορά τη σελίδα 9, δεν είχα χρόνο να το εξετάσω πριν το έγγραφο. Αυτή τη στιγμή το είδαμε. Έτσι λοιπόν, ίσω να μην ε, σα κάνω και τι πλέον κατάλληλε ερωτήσει ούτε πλήρε ερωτήσει, αλλά αν δούμε τα διαγράμματα στην ε, σελίδα 9, βλέπω ότι τα μεγαλύτερα σχέδια έχουν παρουσιαστεί στην προτεραιότητα 3. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αυτό γιατί έγινε, γιατί στην προτεραιότητα 3 από την αρχή έχουν εκταμιευτεί περισσότερα κονδύλια γιατί παρουσιάστηκαν περισσότερα σχέδια. Γιατί πέρα από την προτεραιότητα 3, αυτό που βλέπω εγώ πολύ σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη για το εγγύσμα μέλλον είναι η προτεραιότητα 4. Γιατί εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε αυτές τις λίγες δυνατότητες χρηματοδότησης που έχουμε μέσω ε, και των ιδιωτικών ε, χρηματοδοτήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε μεγάλη έμφαση στην προτεραιότητα 4. Και μια ακόμη ερώτηση για το κόλθο διάγραμμα. Νομίζω ότι σωστό είναι, επικεντρώνεστε εδώ στη συνδρομικό χώρο, αλλά δεν βλέπω πολλά για τις θαλάσσιες μεταφορές. Βλέπω εδώ ε, κάποιες μεταφορές για τις θαλάσσιες οδούς γενικά. Αυτό κατά την άποψή μου είναι μια εναλλακτική μεταφορών, πολύ σημαντική, όμως ε, θα έπρεπε να ενδυναμωθεί λίγο περισσότερο. Και μια τρίτη ερώτηση. Όπως μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Εσείς είπατε ότι υπάρχει και άλλη μία προκήρυξη ε, διαγωνισμού μέχρι τα τέλη του έτους και θα υπάρξει και μία ακόμη προκήρυξη διαγωνισμού ίσως το επόμενο έτος, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, για να καθορίσουμε τις δυνατότητες που έχουμε μέχρι τα τέλη του 2013, σωστά. Δηλαδή από σήμερα μέχρι τα τέλη του 2013, δηλαδή μέχρι το τέλος των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών παραμένουν ένας διαγωνισμός ε, φέτος, μία προκήρυξη φέτος και μία του χρόνου. Θα ήθελα να κατανοήσω κάπως καλύτερα αυτό το προσανατολισμό. Τώρα, να δούμε τις προτάσεις. Βλέπω ότι δεν ε, έχει γίνει ιδιαίτερα σεβαστή αυτή η ανταλλαγή μεταξύ των κρατών ε, εδώ το λαμβάνετε αυτό υπόψη ή απλώς επικεντρώνεστε στα σχέδια. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο μιλητής, ο κ. Αλκαντράουι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, λάβαμε το έγγραφο και μπορούμε να το μελετήσουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να λάβει γέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Καλή φαίνεται η πρόταση εκ πρώτης όψεως και δεν έχω στην πραγματικότητα πρόβλημα με την προτεραιότητα 3. Νομίζω ότι η ιδέα είναι να επενδύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο στο δίκτυο TNT. Ευρωπαϊκά Δίκτυα για τις Μεταφορές. Τώρα, Πρέπει να δούμε και τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις ε, και ξέρω ότι κάποιοι έχουν κατά νου και τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων, όμως ε, νομίζω ότι στο μέλλον αυτό μπορεί να είναι ένα τμήμα του συνολικού μείγματος χρηματοδότησης ε, και θα ξεκολουθούμε να χρειαζόμαστε δημόσια στήριξη, άμεση δημόσια υποστήριξη από τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς για αυτά τα σχέδια, για αυτά τα έργα. Έχω και ένα άλλο σχόλιο που το υποβάλλω κάθε φορά και θα έλεγα ότι σχεδόν ε, το μισό της στήριξης πηγαίνει σε μελέτες. Εμείς θέλουμε όμως να δούμε και πράγματα να υλοποιούνται συγκεκριμένα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσα να σας ρωτήσω αν η εμπειρία σας από τα περασμένα έτη δείχνει ότι μετά από τις μελέτες τελικά έχουμε και υλοποίηση πραγματικών έργων ή θεωρείτε ότι τελματώνουν κάποια σχέδια. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να διερευνήσουμε ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα, ποια ήταν τα πραγματικά αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Όμως κάτι ακόμα. Άκουσα ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή αυτή την εβδομάδα και η ιδέα είναι να καταλήξει σε τελικές αποφάσεις. Ε, θα έρθετε και πάλι σε επαφή με τα κράτη-μέλη και θα τους επιτρέψετε να έχουν ένα τελικό λόγο. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή αυτή η πρόταση είναι τελική, σωστά καταλαβαίνω. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις εξηγήσει και σε σχέση με την πρωτοβουλία που μας έστειλαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν λίγες μέρες. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τη διαδικασία που έχει τεθεί. Καταρχήν, σε αυτή την προκήρυξη βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένα σχέδια που έχουν επιλογή ως προτεραιότητα από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να συμπίπτουν με ορισμένα από τα σχέδια προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί στο Connecting Europe. Επομένω, ε, με ποιο τρόπο θα καταστεί συμβατή αυτή η διαδικασία με την επιλογή αυτών των ε, σχεδίων με την πρωτοβουλία Connecting Europe που με τη σειρά της καθορίζει τα κυρία σχέδια, προσδορίζει τα κυρία σχέδια και θα έχει και μία δυνατότητα χρηματοδότησης. Ε, ε, της αρχής θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να αλληλοεπικαλυφθούν ή αυτή η μελέτη κατά κάποιο τρόπο ε, θα εξυπηρετήσει και το πρόγραμμα Connecting Europe. Δεν κατανοώ ακριβώς πώς θα καταστούν συμβατά αυτά τα δύο εργαλεία, αυτά τα δύο μέσα. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Δεύτερο. Πράγματι, η ανάλυση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και πάλι θα επιστραφεί στην Κομισιόν και αν κατάλαβα καλά, η Κομισιόν θα είναι αυτή που θα αποφασίσει ποια είναι τα σχέδια που θα τυπούν τελικές χρηματοδότησης. Όλα αυτά τα σχέδια και ορισμένα εξ αυτών ε, αφορούν κράτη που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δεινή χρηματοοικονομική και οικονομική κατάσταση και θα απαιτήσετε κάθε κράτος να συνεισφέρει χρηματοοικονομικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν κατά την επιλογή των σχεδίων αυτών αναλύσατε το τμήμα που μπορεί να χρηματοδοτήσει το κάθε κράτος για την εκτέλεση αυτού του έργου. Και τρίτον, Αυτή η επιλογή των ε, σχεδίων θα μπορούσε να απορριφθεί κάποια στιγμή από τα κρατημέλη. Δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Λόγω των ε, περικοπών που μπορεί να υπάρξουν ε, στους προπολογισμούς φέτος και τα επόμενα χρόνια. Έχετε σκεφτεί αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και για το κείμενο που έχουμε δεν μπορώ να τα δω όλα έτσι τώρα στην αρχή. Ορισμένε ερωτήσει όμω. Καταρχά, γιατί φυσικό αέριο και ε, ηλεκτρικέ εθνικέ οδοί, γιατί παίζει ρόλο αυτό. Γενικά μιλάμε για ενέργεια. Και ω Επιτροπή δεν είμαστε αρμόδιοι για αυτό το θέμα τη ενέργεια. Αν κοιτάξω τώρα τους πίνακες, καταλαβαίνω ότι τα ότι σε γενικέ γραμμέ μπορώ να πω ότι, η... ότι προτιμώνται οι σιδηροδρομικές ε, οδοί και όχι ε, οι δρόμοι. Φυσικά αυτό έχει περιβαλλοντική, περιβαλλοντικά προτερήματα, όμως υπάρχει μια αλλαγή, μια προτίμηση προς τους σιδηροδρόμους. σιδηροδρόμους. Αυτό το βρίσκω καλό. Τώρα, όσον αφορά τις ε, πλωτές οδούς, βλέπω ότι έχει μειωθεί η συχνότητα της χρήσης. Τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο δεν βλέπω καμία αναφορά στον Έλβα και στο δούναβη και αυτό θέλω να το καλωσορίσω γιατί είναι πάρα πολύ καλό και εύχομαι να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί, πώς προέκυψε αυτό. Στη Γερμανία οι, μεταφο... οι πλωτές μεταφορές μειώθηκαν ε, στο 18% τον τελευταίο χρόνο και αυτό στο Δούναβι στις εκατομμύρια ευρώ. Το 2000 υπήρχαν 10.000 τόνοι και πέρυσι 6% λιγότερο. Και το να επενδύσει κάποιος πάνω σε αυτό για μένα είναι σπατάλη χρημάτων, άσκοπη. Μετά, τα μέσα των κρατών μελών είναι αποφασιστικό κριτήριο. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που πρέπει να αποφασίσουν. Φυσικά και είναι έργο των εθνικών κοινοβουλίων και των επιτροπών ε, προϋπολογισμού των δημοσιονομικών. Ε, όμως, και βλέποντας όλα αυτά, στη σελίδα 17 για τις ε, σιδηροδρομικές γραμμές. Βλέπω έναν τεράστιο κύκλο γύρω από το Μόναχο, καθοδόν προς το Τωρίνο, και βλέπω ότι όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο κύκλος, τόσο περισσότερα χρήματα πηγαίνουν προς τα εκεί και χρειάζονται. Και αν δούμε Βιέννη Μπρατισλάβα, αυτό το δρομολόγιο, άλλος ένας πάρα πολύ μεγάλος κύκλος, ο διάδρομος προς την Αδριατική, Βαλτική Αδριατική, είναι ένα αυστριακό project το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί και το οποίο έχει εφαρμοστεί για να μην μείνουν απ' έξω κάποιες αυστριακές πόλεις όπως η Klagenfurt για παράδειγμα. Ε, δεν έχει να κάνει αυτό τίποτα με την μεταφορά επιβατών και δικαιολογείται ότι ναι είναι το project Βαλτική Αδριατική και γι' αυτό χρειάζονται κονδύλια όμως από την Πρατισλάβα για να, μέχρι την Αδριατική. Υπάρχει ένα σημείο, ένα ορεινό σημείο που χρειάζονται ε, να ηλεκτροδοτηθούν οι σιδηροδρομικές γραμμές και αυτό κοστίζει φυσικά. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξαναεξετάσουμε αυτά τα μεγάλα project. Το Think Big είναι κάτι που και στο παρελθόν. Πλέον τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Κύριε Ρέτουκ, ε, θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε στα τρία λεπτά. Γιατί όλοι να, μιλά, να μιλάτε παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, βρίσκω το, τις προτάσεις σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Τα περισσότερα από αυτά τα 74 ε, project είναι στην κατηγορία 3, προτεραιότητα 3 στην ολοκλήρωση των τεντή των, ε, σχεδίων TNT. Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι χρηματοδότησης πηγαίνει σε περιβαλλοντικά έργα Δύο project έχουν να κάνουν με την μόλυνση στις ενέργειες και θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά θέλω να ρωτήσω, εδώ μπροστά μας βλέπουμε δέκα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε μια συγκέντρωση των project στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες και ελάχιστα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και μπορείτε να μας πείτε ποιος, λόγο, ποιος είναι ο λόγος. Μετά βλέπω ότι όσον αφορά τη μείωση διοξιδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών. Ε, βλέπω ότι υπάρχει κάποια σάφεια στις, ε, προς, στους ε, διαγωνισμούς. Για ποιο λόγο. Έπειτα. Είναι βέβαια σημαντικό να ολοκληρωθούν αυτά τα τρέχοντα project 10T. Και φυσικά καλώς τονίσατε την, την προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, όσον αφορά την προτεραιότητα 4, έργα δημόσιου ιδιωτικ... δημόσιας ιδιωτικής συνεργασίας, παρατηρώ εδώ, αλλά τι γίνεται με τα χρηματοδοτικά μέσα. Ευχαριστώ. Κύριος Χάουιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κανονικά δεν είμαι μέλος αυτής εδώ της Επιτροπής. Ε, όμως χαίρομαι πάρα πολύ που διάβασα στη σελίδα 100 για την προώθηση των εμπορευματικών μεταφορών μέσω της ε, Μεγάλης Βρετανίας προς την Ιρλανδία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την απόφαση αυτή και σας διαβεβαιώ Έχοντα γνώση του τόπου μου, ότι ε, για μας, για τον τόπο μας, πραγματικά θα δώσει όθηση στην οικονομία, θα επιτρέψει περισσότερο εμπόριο και θα ωφελήσει τις ε, κοινότητες. Ε, κάποιες γρήγορες ερωτήσεις. Πρώτα, ξέρω τη δική την αξία για μας, για τον τόπο μας. Όμως, γιατί υπάρχει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί απασχολεί αυτό την Κομισιόν. Έπειτα από το έγγραφο βλέπω ότι κάποια project είναι έτοιμα να αρχίσουν και θα ήθελα να μάθω πότε αυτά τα project σκοπεύουν να αρχίσουν. Τέλος, ο κ. Πακέ μας περιέγραψε την διαδικασία από εδώ και στο εξής για την Επιτροπή με τα κράτη-μέλη και τις διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Όμως, αν κρίνω από τους προηγούμενους κύκλους διαπραγματεύσεων για τα τέντη, σε ποιο ποσοστό ε, μπορούμε να ε, ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία, τι θα αλλάξει και πόσο θα αλλάξει στην διαδικασία από αυτό το στάδιο στο τελικό στάδιο σύμφωνα με την εμπειρία που έχετε αποκομίσει. Μπορείτε ε, να αναμένετε κάποιες αλλαγές. Ευχαριστώ. Κύριε Μπράντμπορν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρία σύντομα σχόλια. Έριξα μια γρήγορη ματιά στο έγγραφο και μου δημιουργείται η εντύπωση πως αυτή η προσπάθεια που γίνεται για αποσυμφόρηση είναι πολύ σωστή. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε παραπάνω γιατί από τη στιγμή που είναι περιορισμένοι οι πόροι μας νομίζω ότι αυτή είναι και η βέλτιστη χρήση αυτών. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε και η κυρία Μπιλμπάου για την ε, περίπτωση που μπορεί να έχουμε κάποια σύγκρουση με το μέσο Connecting Europe δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε δύο διαφορετικές ε, διαδρομές ή μονοπάτια, γιατί δεν ξέρω αν κάπου θα συναντηθούν ή αν θέλουμε να συναντηθούν. Θα ήθελα λοιπόν να συνταχθώ μαζί της. Τρίτον, για το χρονοδιάγραμμα. Ξέρω πως πολλά από αυτά τα έργα θεωρούνται προτεραιότητες. Αναρωτιέμαι όμως εάν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τη συγχρηματοδότηση των έργων αυτών και θα ήθελα να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν είναι πρόθεσή τους ή αν θα καταθέσουν πρόταση για να έχουν κάποιες ε, ρήτρες ε, sunset clauses ή ε, χρονοδιαγράμματα για το μέχρι πότε μπορούν να ξεκινήσουν αυτά τα έργα ε, έτσι ώστε η χρημοδότηση, ακόμα και η πλασματική που τους έχει κατανεμηθεί να διακόπτεται το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος. Αυτά. Και το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι χαίρομαι για το όσο είπε ο συνάδελφος από την Ανατολική Αγγλία, αλλά πρέπει να σας πω ότι μάλλον παραξενεύομαι γιατί περίμενα και κάποιο σχόλιο για τις βελτιώσεις ή ενδεχόμενες βελτιώσεις από το Φίλιξ μέσω του ε, Α14 και του ε, μη 61 από το Λονδίνο στις βιομηχανικές περιοχές των Midlands. Δεν περιμένω κάποια απάντηση, αλλά ίσως ο κύριος Πακέ θα μπορούσε να δει και αυτή τη σύνδεση, να δούμε αν υποβλήθηκε κάποια πρόταση για την βελτίωση αυτών και κυρίως για την περιοχή των κόμβων ε, ξέρω από τη δική μου εκλογική περιφέρεια πως έχουμε πρόβλημα και συμφόρησης εκεί, αλλά έχουμε και πρόβλημα με πολλά ατυχήματα, γιατί είναι σημείο πολλών ατυχημάτων. Η κυρία Γιάλα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Πακέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε και που σιγά σιγά χωνεύουμε. Ρωτώ, και νομίζω το ίδιο ρώτησαν και οι συνάδελφοι, με ποιο τρόπο σχεδιάζετε εσείς η προκήρυξη αυτή, ο διαγωνισμός αυτός να προσεγγίσει την προετοιμασία των νέων διευρωπαϊκών δικτύων. Τι εννοώ. Αφού ετοιμάζουμε όλα αυτά, αφού έχουμε κάνει την προετοιμασία, έχουμε ε, ετοιμάσει τις βασικές διαδρομές, τους οδικούς άξονες και τους υπόλοιπους άξονες, ε, θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Ξέρω πως κάποια κράτη-μέλη έχουν υποβάλει και μελέτες σκοπιμότητες για το μέλλον. Τι πιστεύετε ότι ε, προτιμούν τα κράτη-μέλη να δουν λίγο το μέλλον μέσα από αυτά τα έργα ή απλώς θα ήθελαν να κλείσουν κάποιες τρύπες του παρελθόντος. Για την πέμπτη προτεραιότητα, για τα διαδρομές ε, για τα εμπορεύματα, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να σχολιάσετε τα όσα σας είπε. Τώρα, προκήρυξη τώρα και άλλες δύο προκήρυξεις διαγωνισμού πριν ε, κλείσει αυτός ο κύκλος, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλό μήνυμα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καταναλώσει τον προϋπολογισμό μας. Γιατί κάθε φορά στην ενδιάμεση αναθεώρηση αυτό που κάνουμε είναι ότι εντάσσουμε ή απεντάσσουμε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα έτσι ώστε αυτοί οι νέοι διαγωνισμοί να είναι προφανώς ότι έγιναν γιατί κάναμε μια απογραφή και λάβαμε υπόψη τα διδάγματα. Ε, για τα κράτη της νέας συνοχής. Είδα ότι έχουμε έργα στην Πολωνία, στις χώρες Βαλτικής. Μπορείτε να μας πείτε αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να μην έχουμε πλέον επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο στο μέλλον. Να δούμε πώς μπορούν αυτά που μάθαμε να εφαρμοστούν και στο μέλλον. Γιατί σκέφτομαι ακόμα αυτά τα δέκα δις. Έχουμε πολλούς ε, ε, ετούντες οι οποίοι να μην προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Δηλαδή να δούμε πώς χωρίζεται οι αιτήσει ιδιωτικού και δημόσιου. Ο κ. Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, κύριο Πακέ και την Επιτροπή για την παρουσίαση σήμερα των ε, σχεδίων που έχουν εγκριθεί, που έχουν επιλεγεί. Δύο μόνο ερωτήσεις γιατί ήδη τα περισσότερα θέματα έχουν εθιγεί η μία είναι το γεγονός ότι αυτά τα σχέδια βρίσκονται σε μία περίοδο μετέχμιο από τις, την παλιά λογική, την μέχρι τώρα ισχύουσα λογική στα διευρωπαϊκά δίκτυα και λίγο πριν, όπως όλοι ελπίζουμε, την εφαρμογή της νέας περίοδου. Πώς αυτό επηρεάζεται και πώς μπορεί να γίνει η σωστή διασύνδεση των δύο διαφορετικών αυτών περιόδων εφαρμογής της ίδιας στρατηγικής. Αλλά δύο διαφορετικές, έχουμε δύο διαφορετικές περιόδους. Και το δεύτερο είναι, αφορά τα ομόλογα έργου. Και η ερώτηση είναι αν τα ομόλογα έργου που βρίσκονται ήδη, αποφασίστηκε η πιλωτική τους φάση και λειτουργία, θα επηρεάσουν ή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ή μπορούν να βοηθήσουν την υλοποίηση των έργων για τα οποία συζητάμε σήμερα. Mrs. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω πολλά, τα είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Βρίσκω όμω πολύ καλό όλο το κείμενο. Ο κύριος Παρκείδη μας το παρουσίασε και, μας είπε, και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο διακρατικό, αλλά και διατομεακό. Πέρα από αυτά, με, ενδιαφέρε, πάρα πολύ αυτό που είπε ο κύριος Κουμουτσάκο με τα ομόλογα έργου. Θεωρώ πάρα πολύ, σημαντικό, ε, πολύ σημαντική αυτή την παρατήρηση. Υπάρχουν 230 εκατομμύρια κονδύλια που ε, θα χρησιμοποιηθούν και καλό θα είναι να υπάρχει ένας κατάλογος με ποια ε, project θα πάρουν πόσα κονδύλια. Έπειτα πιστεύω ότι η αρχή του use it or lose it, χρησιμοποίησε το ή χάστο, ε, είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και σε αυτά τα project. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, Ρικέ. Κύριος Ρικέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν και τον κύριο Πακέ για την παρουσίαση του εγγράφου. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει και δύο σχόλια. πρώτη παρατήρηση είναι εξή. Εγώ κατανοώ ότι στα πλαίσια του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου είχαμε ένα γνωστό μηχανισμό και συνεχίζουμε. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν έχουμε ένα εκατομμύριο στις προοπτικές. Αλλά δεν είναι το πραγματικότητα όμως το δεύτερο παρατήρηση είναι ότι ακριβώς αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε την ε, σπανιότητα των ε, έργων στις χώρες της συνοχής και πρέπει να υπογραμμίσω πόσο απαραίτητο είναι στην περίπτωση των νοσκοτηρίων να έχουμε 10 ε, δισεκατομμύρια για τις χώρες της συνοχής για να συμμετέχουν στα προγράμματα των ευρωπαϊκών δικτύων. Αλλά έχω και δύο ερωτήσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα το πρόγραμμα θα εξαντληθεί στο χαρτοφυλάκιο που έχουμε σήμερα και που ε, ανταποκρίνεται στο σχέδιο στα σχέδια που έχουμε στη μελέτη σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι εξή. Προφανώ δεν μπορείτε ε, δεν ε, μπορείτε ε, να βάλετε σε αυτό το είδους το πρόγραμμα τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν δετηθούν από τα ομόλογα έργου, αλλά έχουμε του χρηματοδοτικού οργανισμού. συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το χαρτοφυλάκιο που προτείνεται και μπορούν ε, αυτοί οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να τα χρησιμοποιήσουν, ερωτηματικό. Και σκέφτεστε ε, ότι το γεγονός ε, ότι αλλάζεται δημοσιονομικό όγκο στα πλούσια των πολιτών στο δημοσιονομικό προοπτικών θα σας ε, ε, οδηγήσει στο να περάσετε σε λιγότερες μελέτες και σε περισσότερα έργα. Ο κύριος Λιμπεράτς. Ευχαριστώ. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον ε, το κείμενο και τις προτάσεις και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ε, από ό,τι είδα θα υπάρχουν συνολικά 37 εκατομμύρια επενδύσεων στην Πολωνία και τις κατασκευές και 2,7 εκατομμύρια για μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι η πολωνική κυβέρνηση ζήτησε ε, αυτό το ποσό, ένα τμήμα, ένα ποσό απορρίφθηκε, αλλά αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω κι εγώ κάτι κύριε Πακέ. Καταρχήν ε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση του εγγράφου αυτού και εγώ έριξα μια γρήγορη ματιά και πραγματικά με εξέπληξε, όπως και άλλους συναδελφούς, ο τρόπος που όχι μόνο προσπαθείτε να συνδέσετε τις προτεραιότητες με το διασυνοριακή συνιστόσα, που είναι μια προτεραιότητα που έχει θέσει πάντοτε αυτή η Επιτροπή, αλλά με εξέπληξε και το γεγονός ότι προσπαθήσατε το να υπάρχει και διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφορών και να διασφαλίσετε ότι εκεί όπου έχουμε ε, διευρωπαϊκά δίκτυα συνεχίζονται και εκεί τα έργα για να υπάρξουν βελτιώσεις. Έτσι λοιπόν συνολικά νομίζω ότι είναι καλό το έγγραφο από όσο κατανοώ τώρα θα σταλούν στα κράτη-μέλη, αλλά για να απαντήσω εγώ κατά κάποιο τρόπο πριν από εσάς τον κύριο Χάουιτ, είναι πολύ σπάνιο να γίνουν αλλαγές σε αυτό, το έγγραφο, σε αυτό το έγγραφο και αν γίνουν θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί. Έτσι λοιπόν εγώ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και ριζοσπαστικά αλλά μάλλον θα το επιβεβαιώσει αυτό και ο κύριος Πακέ όταν θα απαντήσει στην ερώτησή σας. Παρακαλώ, κύριε Πακέ, έχετε πολλά να απαντήσετε. Από πού θα ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ξεχάσω πολλά και αν ε, ξεχάσω σας ζητώ ίδιο συγγνώμη, αλλά βάσει των σημειώσεων θα σας απαντήσω γραπτός. Για να ομοδοποιήσω ορισμένα από τα σχόλια, ίσως να επανέλθω στη διαδικασία και να πω ότι όλα αυτά τα project ε, τα οποία είναι στη σύσταση παρουσιάστηκαν από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή κανένα από αυτά τα σχεδία δεν ε, έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένα από την Κομισιόν ή από την υπηρεσία ή από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες πάντοτε ο δικαιούχο είναι αυτό που ζητά τη χρηματοδότηση και στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη, και αυτό ήταν σημαντικό σημείο τη αξιολόγηση, έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι η χρηματοδότηση θα ήταν διαθέσιμη. Και ένα στοιχείο του κριτηρίου της οριμότητας είναι να δούμε αν υπάρχει ε, στέρεα χρηματοδότηση και αν μπορεί να εφαρμοστεί η ε, συμμετοχή έτσι όπως παρουσιάζεται στην πρόταση. Ο κ. σε αυτό το θέμα μάλιστα. Και ελεγχθέντως αυτού οι προτάσεις. Νομίζω ότι δόθηκαν φέτος τον Απρίλιο και τώρα θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις χρηματοδότησης πριν τα τέλη του έτους και τα 74 σχέδια αν επιβεβαιωθούν από την Επιτροπή των Κρατών Μελών αυτή την εβδομάδα και φυσικά αν δούμε και είναι και εμπειρία των προηγούμενων ετών αλλά δεδομένου ότι έχει γίνει εκτεμίευση του συνολικού προπολογισμού, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών και η πραγματικότητα τα τελευταία πέντε έτη είναι ότι τα κράτη-μέλη γενικά υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν ως έχει. Αυτό είναι λοιπόν ένα πιθανό σενάριο για τη συνάντηση της Πέμπτης. Έτσι λοιπόν, κατόπιν ξανασυζητούνται αυτές οι 74 προτάσεις με τα κράτη-μέλη. Αυτό γίνεται από τον οργανισμό και λαμβάνεται, μάλλον και προετοιμάζεται μια συγκεκριμένη απόφαση χρηματοδότησης και φυσικά στο κάνουμε αυτό θα ξαναεξετάσουμε το θέμα της χρηματοδότησης, θα ξανατεθεί αυτό το ερώτημα, δηλαδή είπατε ότι θα κάνετε αυτό, ε, ήταν πιστικό, εμείς θα χρηματοδοτήσουμε την πλευρά μας, εσείς μπορείτε να χρηματοδοτήσετε, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Και επίση το Use it or lose it θα συνεχίσει να ισχύει. Είναι μία από τις αρχές ε, του προγράμματος ε, ΔΕΔ για μεταφορές και φυσικά θα ε, πρέπει να προωθεί και να εφαρμοστεί. Αλλά το θέμα της χρηματοδότησης είναι φυσικά μία ενισχύα και για την Κομισιόν υπό τις σημερινές συνθήκες και για τους μηχανισμούς του προγράμματος και στο στάδιο της επιλογής και στο στάδιο της εφαρμογής. Όλα αυτά είναι υπό έλεγχο θα υπάρξουν άλλες προκήρυξεις διαγωνισμού, όπως είπα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υπάρχει μια προκήρυξη διαγωνισμού για τα έργα προτεραιότητας. Αυτή η ετήσια προκήρυξη διαγωνισμού δεν είχε επικεντρωθεί σε εκείνα τα σχέδια. Αυτή που θα εμφανιστεί το 2012 θα επικεντρώνεται σε αυτά τα project προτεραιότητας ε, και αυτό που θα δούμε το 2013 θα είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα, σύμφωνα με αυτό που εξετάζεται σήμερα το απόγευμα, αλλά θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι ορισμένα από τα σχολεία σας ίσως ε, να ε, μας οθούν να το σκεφτούμε λίγο παρατέρω πριν να το παρουσιάσουμε, αλλά θα έχουμε όπως και να έχει δύο ε, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και υπάρχει μια δυνατότητα να έχουμε μια τελευταία προκήρυξη το 2013 η κυρία Αγιάλα, αν δούμε ότι παραμένουν κονδύλια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των κονδυλίων, μπορούμε να έχουμε μια νέα προκήρυξη διαγωνισμού το 2013, ανάλογα με τι επιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων που θα μπορούσαν να διατεθούν από αυτά τα project. Το σημαντικό είναι τώρα να έχουμε το 2012 ε, μια προκήρυξη για τα σχέδια προτεραιότητα, πολυετή προκήρυξη και θα έχουμε και άλλο ένα διαγωνισμό το 2013 στι αρχέ εχουμε Έχουμε γράψει αυτά ποσά 3 2-3-4 φορές, έτσι λοιπόν δεν έχω ανησυχία ότι θα χρησιμοποιηθεί ο προπολογισμό και το 2012 και το 2013, αλλά και ο συνολικός προπολογισμό του προγράμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι διάφορε συνιστώσει και προτεραιότητες ε, στην προκήρυξη, θέλω να ευχαριστήσω τα βουλευτέ για τα σχόλιά του. Να πω ότι και εγώ θα ήθελα να δω περισσότερα για τις πλωτές οδούς, για τις θαλάσσιες μεταφορές και αντικατοπτρίζεται ε, ένα μικρότερο μερίδιο ε, για αυτά τα project σε σχέση με το τι παρουσιάζεται είναι καλής ποιότητας. Έτσι λοιπόν έχουμε λιγότερα project και επίσης ε, στο σιδηρόδρομο χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, όμως έχουμε όλο ένα και καλύτερης ποιότητας project για τις ε, πλωτές μεταφορές, όχι τόσο για το Δούναβι και για τον Ελβα, αλλά στις χώρες Μπενελούξ περισσότερο κεντρωνόμαστε. και τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πού θα ζητήσουν χρηματοδότηση και φέτος ε, αυτά τα σχέδια ήταν όνομα και θεωρήθηκε η συγχρηματοδότηση χρήσιμη. Και σαφώς οι προτεραιότητες του ίδιου του προγράμματος εργασίας. Δηλαδή αυτές που θέσατε όταν εμείς ε, ε, δημοσίευσαμε την κρίξη είχαν να κάνουν με του σιδηροδρόμους και με τις πλωτές μεταφορές, ενώ οι οδικές μεταφορές ε, ήταν περισσότερο στο περιθώριο. Και αυτό εξηγεί και γιατί έχουμε λιγότερα project σε αυτό το τομέα. Τώρα υπάρχει και το ερώτημα για τη σύνδεση μεταξύ του μέσου Connecting Europe και αυτού του εγχειρήματο ως ε, ένα βαθμό αναφέρθηκε σε αυτό το Ε, Αυτό το ετήσιο πρόγραμμα βασίζεται στις εφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, ε, στα εφιστάμενο πρόγραμμα ε, δέντια για τις μεταφορές. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι με αυτό το τελευταίο στάδιο του προγράμματος TNT θα έχουμε και μια γέφυρα για το μέσο Connecting Room και για το νέο πρόγραμμα TNT. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις διάφορες προτάσεις, ένα μεγάλος αριθμός προτάσεων που επίση επίσης το παράτημα ε, του μέσου της διασύνδεσης για την Ευρώπη και φυσικά αυτό θα καταστεί ακόμη πιο ορατό, πιο προφανές στο πολιτές ε, πρόγραμμα. Αργότερα φέτος θα επικεντρωθούμε ε, σε σχέδια που είναι τώρα στο δίκτυο γιατί τώρα έχουμε τη διαδικασία συναπόφασης εκεί αλλά υπάρχει ήδη ένα σύνδεσμο. Φυσικά θα υπάρχουν και κάποια σχέδια που θα εφαρμοστούν από μόνα του. Ελπίζουμε ότι θα συμπληρωθούν με τη χρηματοδότηση που προβλέπετε εδώ και αν όχι θα ολοκληρωθούν δυνάμει των προκηρύξεων του 2013 ή από πόρους των κρατών ή βάση άλλων προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από τον προβληματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει να βρούμε ένα μεγαλύτερο συνδεσμό με το μέσο Connecting Europe και το κάνουμε αυτό με περισσότερε προτεραιότητε στον τομέα των μεταφορών, με την καινοτομία, με τι καθαρέ μεταφορέ. Δικαιοτοπίζεται αυτό στο Connecting Europe Facility και ε, στο δέντρο για τι μεταφορέ, αλλά πιο συγκεκριμένα με την προτεραιότητα 3. Φυσικά στο στάδιο τη μελέτη για τι προτεραιότητα 3. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παρουσιάσω αριθμητικά στοιχεία, αλλά πολλές από αυτές τις μελέτες στη συνέχεια οδηγούν σε project, γιατί όταν μιλάμε για μελέτες, για τον τι έχετε φυσικά και μελέτε μελέτες σκοπιμότητας, αλλά περισσότερα χρήματα, τα περισσότερα χρήματα της μελέτες πηγαίνουν στις μελλοντικές, στις ε, ε, περιβαλλοντικές μελέτες αντικτύπου ή σε διερευνητικές μελέτες που σχετίζονται σε, με συγκεκριμένο έργο τεντή στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, μια μελέτη στη συνέχεια μεταφράζεται σε σχέδιο τεντή και ίσως εδώ μπορεί να γίνει και ο σύνδεσμος ε, πιο στενά με το Connecting Europe. Δηλαδή, ελπίζουμε να χρησιμοποιηθεί η προτεραιότητα 3 από τα κράτη-μέλη για να προετοιμάσουν το κατάλογο στο παράρτημα τη πρόταση τη Κομισιόν. Αλλά, όπω σωστά τονίστηκε, Λίγα μελη νέα κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα και νομίζω ότι για το τελευταίο ετήσιο πρόγραμμα πρέπει να δούμε αν θα υπάρχει πιο συγκεκριμένο σύνδεσμο τη προτεραιότητα 3 με το παράρτημα. Η δυσκολία είναι πρόταση της Κομισιόν ε, και κάποια στιγμή θα συμμετέχετε κι εσείς και στο Συμβούλιο στη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε ότι η ε, εναπομείνασα χρηματοδότηση θα προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος για το μέσο Connecting Europe. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να είναι ενημερωμένα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Και το τελευταίο γενικό μου σχόλιο είναι για το ομολογάριο για την προτεραιότητα 4 και για την καινοτόμο χρηματοδότηση. Τα σχέδια στην προτεραιότητα 4 νομίζω είναι 6 Πρόκειται για μελέτε που θα, βοηθήσουν τους Δικαιούχου ε, να αξιολογήσουν πόσο, πόσο μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα όπου θα ε, χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση περισσότερα από αυτά τα έργα, στα πλαίσια των ε, έργων αυτών θα μπορούσε να αποφασιστεί πότε έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και πότε οι παράμετροι ε, της θα πληρούνται και μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια το ομόλογα έργο. Έτσι λοιπόν προετοιμάζουν το έδαφος για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ομόλογα έργου. Μόνο έξι σχέδια έχουμε στο στάδιο αυτό. Νομίζω ότι έχουμε τα διπλά από πέρσι. Καλή είναι η τάση. Λοιπόν, βέβαια εξακολουθεί να είναι μικρό ο ρυθμός, έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι εδώ η δουλειά για το αποθεματικό σχεδίων θα μας ε, οδηγήσει σε περισσότερη γνώση και θα έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση για χρηματοδότηση τα επόμενα έτη ή στο επόμενο ετήσιο πρόγραμμα. Νομίζω ότι με αυτά κάλυψα τις περισσότερες ε, οριζόντιες ερωτήσεις να φερθώ και στα υπόλοιπα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Νομίζω πως μένουν μόνο τα σχόλια του κυρίου Κράμερ δεν είναι Βαλτική Αδριατική, όμως τώρα είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε να κοιτάξετε τις λεπτομέρειες του project. Είναι ένα πολύ μικρότερη εμβέλεια έργο. Εάν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις, τα μεγάλα έργα υποδομής, είναι διαφορετικό στο ΣΕΦ και όχι σε αυτό εδώ. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Χιουίτ για τα σχόλια του σχετικά με τα με το project που συνδέει το Show με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του, της σύνδεσης των ΣΕΦ και των ε, ΤΕΝΤΗ, της σύνδεσης των ευρωπαϊκών λιμένων με, τα, ε, με την εσωτερική, ε, με την ενδοχώρα και είναι στο χέρι και των κρατών μελών και, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παραδώσουν περισσότερο λειτουργικές ε, χρήσεις των δικτύων αυτών. Νομίζω πως ε, απάντησα τα περισσότερα σχόλια, αλλά θα επανέλθω και θα απαντήσω στα σχόλια του κυρίου Μπράντμπερν για την περιοχή Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Και νομίζω ότι τώρα έχω καλύψει αυτά που ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρκέ, για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών. Τώρα Αναμένουμε την απόφαση της Πέμπτης από τα κρατημέλη και μετά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το γρηγορότερο δυνατόν να πάρουμε τα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί στα έργα αυτά που το χρειάζονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δεν νομίζω να σας ξαναδούμε πριν τις διακοπές, οπότε καλά να περάσετε. Θα σας δούμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Κύριε Γκρίσμπεκ, Κύριε Γκρίσπεκ, η κυρία Γκρίσπεκ ε, με ενημέρωσε ότι θα τρέχει από αίθουσα σε αίθουσα γιατί είναι και, στην, ε, και σε άλλη επιτροπή, στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων τώρα. Ορίζοντας 2020 η Ήτρα είναι η αρμόδια επιτροπή. Η κυρία Γκρίσπεκ θα έχει συντάξει την έκθεση, έχετε το λόγο κυρία Γκρίσμπεκ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα να σας παρουσιάζω αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης Horizon 2020 και να σας ευχηθώ καλή συνεργασία για τις επόμενες εβδομάδες. Ακόμα και αν αυτές οι εβδομάδες θα αφιερωθούν πιο πολύ στη χαλάρωση. Πριν μπω στα θέματα ουσίας, θα ήθελα επί της διαδικασίας να κάνω το εξής σχόλιο. Δύο έγγραφα ήρθαν στην Επιτροπή μας. Έχουμε τον κανονισμό 809, πρόγραμμα πλαίσιο, συναπόφαση και το 811 ειδικά προγράμματα που είναι σύμφωνα με τη διαδικασία της διαβούλευσης. Εκεί είναι περιορισμένος ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Αποφάσισα λοιπόν να σας προτείνω να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο πρόγραμμα πλαίσιο με κάποια στοιχεία τα οποία θα σας φανούν πιο σημαντικά από τα ειδικά προγράμματα, να τα εντάξουμε και αυτά μέσω των τροπολογιών. Για να δούμε την ουσία του θέματος και πριν μπούμε στις λεπτομέρειες του Horizon 2020, να σας πω πως είναι τα κλειδιά του παραδείσου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έρευνα, για την καινοτομία. Όλοι εξυπηρετούμε τους ίδιους στόχους και σε μια στιγμή χρονική όπου η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε εκεί όλες μας προσπάθειες. Θα πρέπει σε πολλούς κλάδους εδώ στην Ευρώπη να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί να είμαστε πιο ισχυροί από τα τρίτα κράτη και νομίζω πως τα νέα στοιχεία σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση σημαίνουν πως η ήπειρός μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενορχιστρώσει αυτές τις βαθιές αλλαγές που χρειάζονται για να στηρίξουν τις οικονομίες, για να προχωρήσουμε στην έρευνα και την τεχνολογία, για να γίνουμε σε βιομηχανικό επίπεδο πιο ανταγωνιστικοί. Αυτή λοιπόν η έκθεση Horizon 2020 θέλει να εξασφαλίσει τη δική μας βιομηχανική κυριαρχία επί του κόσμου και να είμαστε σε επιστημονικό εθνικό επίπεδο η άριστη. Μεταφορές, μεταφορές στον πληθυντικό, κομβικός κλάδος της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να γίνουμε πιο ολοκληρωμένοι, να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε και κάποιες κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι μία με την οποία μπορώ να συνταχθώ απόλυτα, ότι δηλαδή κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο εγκρίνω πριν από μερικού μήνε, ε, την έκθεση Gross για την ενιαία Ευρώπη των μεταφορών και πιστεύω πως θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την ε, κατεύθυνση. Θα αναφερθώ σε μια βασική πτυχή της πολιτικής μεταφορών που είναι το θέμα της ενέργειας και της επιπτώσεις που έχουν οι μεταφορές στην κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιούμε για τις μεταφορές, γιατί τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι αιώνια και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον υπερβολικά μεγάλες. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα της εξάρτησης από αυτά. Οι εκπομπές και οι οροφές των εκπομπών, ανάλογα με το μέσο συγκοινωνίας, θα αποφασιστούν 3-20, είπαμε 3 επί 20, Έχουμε στην έκθεση τους, στόχου ε, στόχους 2020, το 3 επί 20 λοιπόν το πολλαπλασιάσαμε και μπορώ να σας πω θα κάνουμε τις διορθώσεις. Για να τα πετύχουμε πρέπει λοιπόν οι μπαταρίες, οι κινητήρες, οι υποδομές μας να γίνουν πιο ε, καινοτόμες, να εξοικονομούν ενέργεια και να δούμε αν θα βρούμε κάποια καύσιμα υποκατάστατα που θα είναι βιώσιμα. Αυτά θα συνδυάζονται με μια στρατηγική διαχείριση αποβλήτων και προ την ίδια κατεύθυνση προτείνω σε στενή συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε και τον αεροδυναμικό σχεδιασμό των οχημάτων, κάτι το οποίο θα βελτιώσει τις επιδόσεις του, του κόσμου των μεταφορών. Δηλαδή μιλάμε για ευφυείς μεταφορές. Το άλλο που είδαμε είναι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ανάγκη της κινητικότητας που αυξάνεται μαζί με την ελεύθερη ροή της συγκοινωνίας. Φτάνοντας σε ένα σύστημα πολυμεσικό, προσβάσιμο, ε, συνεκτικό, σε υποδομές καινοτόμες, ποιοτικέ που θα χρησιμοποιούν όλα τα μέσα. Θα πρέπει οι των Ευρωπαίων μια και τα ενδιατήματά τους εξελίσσονται στην Ευρώπη, θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις κομβικές πτυχές. Και να δούμε ποια θα είναι η κινητικότητα στις αστικές περιοχές. Αυτή είναι η βασική μας πρόκληση. Είναι μια πρόκληση οικονομική, είναι πρόκληση για την απασχόληση, αλλά επίσης είναι πρόκληση και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων ε, στα αστικά, στις αστικές ζώνες. Προτείνω λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ε, την βιωσιμότητα και τις κοινωνικές ε, ανάγκες τη στιγμή του σχεδιασμού αυτών των νέων μεταφορικών μέσων, έτσι ώστε να εξαλείψουμε την ανισότητα και να βελτιώσουμε την κατάσταση των χρηστών, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Στα πλαίσια αυτά, η δημιουργία της κοινότητας της γνώσης και της κοινοτομίας για την αστική κοινοτικότητα είναι το καλύτερο και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Έτσι λοιπόν εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα έρευνας, στα πλαίσια των όσων κάνουμε, στο κέντρο των όσων κάνουμε θα πρέπει να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε την βιώσιμη κινητικότητα ε, χρησιμοποιώντας ε, τις πιο καινοτόμες λύσεις για την μετακίνηση εμπορευμάτων ε, και επιβατών έτσι ώστε να μειώσουμε τη ρήπανση, την ηχορύπανση αλλά και για να μπορούμε να προμηθεύουμε πάντα τις αγορές μας. Κοιτάξτε, η αύξηση της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και οι αυξήσει των μεταφορών και όλες οι κατευθύνσεις που σας έδειξα στην αρχή θα πρέπει να μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε αλλά και να τονίσουμε την πτυχή της ανάπτυξης της καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στον κλάδο των μεταφορών για να ε, ε, ξαναξεκινήσει η ανάπτυξη για να ανακάμψουν οι οικονομίες μας και οι κοινωνίες μας, να χρησιμοποιήσουμε τις ευφυείς μεταφορές, το είδατε κι εσείς. Αυτές είναι οι επιταγές στις οποίες θα πρέπει να υπηρετήσει η Ευρώπη για κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς λόγους. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μπορέσετε να συμφωνήσετε μαζί μου και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τη γνωμοδότηση αυτή για τον ρίσο του 2020. Καταρχήν θα να σας πω ότι στη σημερινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προσπαθούμε ε, να σχεδιάσουμε κάποια ευφύ συστήματα μεταφορών. Έτσι λοιπόν από την σκοπιά της Επιτροπής μας πρέπει να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών που θα είναι φιλικό προς τους χρήστες αλλά και προς το περιβάλλον. Οι μεταφορές και οι ε, παραγωγή εξοπλισμού αποτελούν το 6,3% του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό υπάρχει ανταγωνισμός σε άλλα τμήματα του πλανήτη και θα πρέπει τώρα να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να μετριάσουμε ε, τα μειονεκτήματα του σημερινού συστήματος, ε, το να εισαγάγουμε νέες ε, λύσεις και με καινοτόμα τεχνολογία για τη διαχείριση των μεταφορών προκειμένου να έχουμε ένα πιο καθαρό σύστημα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί πολλές επενδύσεις και η λύση θα μπορούσε να δοθεί μέσα από τον οριζόντα 2020. Θα πρέπει ο τομέα να περιορίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να μην εξαρτώμαστε τόσο από το πετρέλαιο, διατηρώντα ταυτόχρονα υψηλή κινητικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει με μια αλλαγή ριζική στα συστήματα μεταφορών και με καινοτόμα συστήματα, εφαρμόζοντας κάποιες ευφυείς λύσεις. Ο τομέας των μεταφορών είναι το μέσο κλειδί γιατί εγγυάται την κινητικότητα των ανθρώπων και των αγαθών. Το σύστημα μεταφορών προσφέρει μία από τις μεγαλύτερες αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Έτσι λοιπόν η χρηματοδότηση της καινοτομίας στον χώρο των μεταφορών θα συμπληρώσει τις δράσεις των κατορμελών. Μία σωστή εφαρμογή του προγράμματος ορίζοντας 2020 θα υποστηρίξει δράσεις που έχουν διευκρινιστεί στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές δράσεις για να αναπτυχθεί ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών η ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών θα συνεισφέρει στην εφαρμογή των πολιτικών στόχων που αναφέρονται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως η βιομηχανική πολιτική ε, σε μια ε, παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη ή στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Κυρία Γιάλη για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Γκρίσπεκ. Ε, επίσης χαίρομαι που μπορώ να συνεργαστώ μαζί της για την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Και ε, εγώ θεωρώ πολύ σημαντικά το όσα υπογράμμισε συνάδελφος, αλλά και την αναγκαιότητα να λάβουμε υπόψη και στοιχεία όπως η ασφάλεια, η καινοτομία ε, μεταξύ χρήστη, οχήματος και υποδομής. Αυτό συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό και στην περίπτωση των ε, οδηγών. Είδαμε και εκεί σημαντικά στοιχεία. Επίσης, το θέμα της κοινωνικής συμπεριφοράς ε, βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κάποιες ομάδες, οι νέοι, τα παιδιά να ε, ε, είναι ομάδες όπου πρέπει να εστιάσουμε σε σχέση με την ασφάλεια. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε και από αυτού και επίσης έχουμε το θέμα της επιμελητίας το ανέφερε η και την υποστηρίζω στην και όταν εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα της ε, οργάνωσης ε, και ε, σε επίπεδο πόλης και στο πώς συνεπάρχουν οι άνθρωποι στην πόλη, πώς συνεπάρχουν οι πολίτες και πώς γίνεται η προμήθεια των αγαθών που χρειάζονται. Τώρα να έχουμε ένα καινοτόμο δίκτυο προμηθειών, το είδαμε αυτό, έχουμε και τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, ξέρουμε πώς πρέπει να τα τροφοδοτήσουμε, όμως σε επίπεδο πόλεων υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να εντοπίσουμε αυτές τις δυσκολίες και να βρούμε καινοτόμως λύσεις. Τώρα για τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι στα χρηματοδοτικά μέσα το είδαμε, αλλά και στην έρευνα Είδαμε πώς έχουμε προσαρμογή νέων τρόπων χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία έρευνα κοινωνικο-οικονομική. Πολλές φορές δεν λαμβάνονται ε, υπόψη γιατί πολλές φορές ε, μιλάμε για έρευνα ε, στο εργαστήριο με το σωλήνα. Όμως υπάρχουν και κάποιες σε ό,τι αφορά τώρα το παγκόσμιο χαρακτήρα, το καθαλικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι είπαμε πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται σε ό,τι αφορά ε, τι συμβάσει σε καθολικό επίπεδο. Δηλαδή πολλές φορές δεχόμαστε να έχει κάποιο ηγετική θέση χωρίς όμως ε, να έχουμε υποστημονικά στοιχεία και επίσης για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Όταν ε, ρωτάμε την Επιτροπή, όταν δημιουργούμε αυτές τις νέες αγορές με τα καινοτόμα στοιχεία της κινητικότητας, της μείωσης του δεξιδιού του άνθρακα κτλ, δεν ε, μπορούμε να έχουμε αριθμητικά στοιχεία για τις θέσεις εργασία που από τη μία χάνονται, από την άλλη κερδίζονται. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εργαστούμε επί αυτής της αξιολόγησης της κοινωνικο-οικονομικής και όταν υπάρχουν αξίες σε σχέση με τις ε, δημόσιες υπηρεσίες για την ασφάλεια, για την ποιότητά του, τους. Ε, νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει επαρκής έρευνα για να δούμε πώς εφαρμόζονται στις δημόσιες υπηρεσίες αυτές οι πτυχές της ποιότητας κτλ. Και σε ό,τι αφορά το κοινωνικονομικό τομέα έχουμε δει κάποιες συγκρούσεις, αλλά τώρα με τις νέες υποδομές, με τα νέα δίκτυα υποδομών πρέπει να δούμε πώς αντιδρούν κάθε φορά οι πολίτες ε, ε, όταν ανακοινώνονται νέες υποδομές. Εγώ νομίζω ότι εδώ η Επιτροπή θα έπρεπε να εργαστεί ε, μέσω της κοινωνικονομική έρευνας για να δει πώς θα επιλύσει αυτές τις κοινωνικές συγκρούσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Ντύρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έργο της. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις ε, κύριες γραμμές που παρουσίασε. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω κάποια συμπληρωματικά στοιχεία Πιστεύω ότι σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, πρέπει να τονίσουμε κυρίως το θέμα της προσφοράς ε, των μεταφορών, ε, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε και στο θέμα της ζήτησης. Δηλαδή όχι μόνο να επιμένουμε στις υποδομές ή στις αποδοτικές μεταφορές, αλλά πρέπει να επιμένουμε και στο πώς θα αλλάξει η συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και των οντολοδοτών. Ε, το 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι συγκεντρωμένο στις πόλεις, έτσι λοιπόν πρέπει αυτό να το λεβούμε υπόψη και θα πρέπει να εργαστούμε εκεί στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά θα πρέπει να δούμε και τη δημιουργία των θέσεων εργασίας και ε, αν ε, όλος ο τομέας των μεταφορών, των αστικών μεταφορών μπορούν να δημιουργήσουν ε, και κάποιες ε, συνθήκες βελτίωσης της διαβίωσης ε, των ανθρώπων που ζουν στην πόλη. Όπως χωροταξία, παραδείγματος χάρη, και κατόπιν θα ήθελα να τονίσω το σύνδεσμο μεταξύ της, των ασφαλών μεταφορών αλλά και των συνδικών εργασίας του προσωπικού. νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και στο πρόγραμμα πλαίσιο και επίσης σε σχέση ε, με ε, την ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Έχουμε δηλαδή τρία συγκεκριμένα συμπληρωματικά στοιχεία όπου θα μπορούσα να κάνω κάποιες ε, τροπολογίες για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές προτάσεις για συγκεκριμένα σχέδια. Ο κύριος Νταμιάννη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να σχολιάσω τα λεγόμενα σας. Καταρχάς να πω ότι για εμείς καλωσορίζουμε την έκθεση της κυρίας Γκρίσπεκ. Ε, διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση σε, ανάμεσα σε αυτήν την έκθεση και σε αυτά που προτείνει ο ορίζοντας 2020. Και αυτό εμπνέει, ε, είναι, έμπνευση για, την, ε, για τις μεταφορές και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η συμφιλίωση της, ε, των στόχων της πολιτικής και της ανταγωνιστικότητας, ο, το φόκους της προκλήσεις στις ενεργειακές, στις περιβαλλοντικές, στις κλιματικές, αυτή η ολιστική προσέγγιση του να βλέπουμε τις μεταφορές ως ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα είναι ένας μεγάλος στόχος η έμφαση στην καινοτομία, η, η προσοχή στις και η έμφαση στις καινοτόμες λύσεις, στις επιπτώσεις στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας. Επίσης, καλωσορίζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ιδιαίτερη έμφαση που η συγγήτρια έχει δώσει σε ορισμένες συγκεκριμένες απόψεις στις πηγές ενέργειας, στις επιπτώσεις στην υγεία, στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και, και μεγαλύτερη έμφαση στις αστικές μεταφορές, στην, στην σύνδεση μαζί με άλλες πρωτοβουλίες στα πλαίσια του Connecting Europe. Υπάρχουν μόνο λίγες Τη της έκθεση αυτής και των ε, τροπολογιών που έχουν προταθεί, που εμείς θα θέλαμε ίσως να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση ή πάνω στις οποίες διατυπώνουμε ορισμένε ανησυχίες. Θα σας πω λίγα παραδείγματα. Ε, τροπολογίες 18 έως 20 για, το, για τη διεπιφάνεια των του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Ε, αυτό, με αυτό ασχολείται ένα άλλο μέρος του προγράμματος και πρέπει να προσέξουμε να υπάρξει ένας ευθύς ε, του τι καλύπτουμε εκεί και του τι καλύπτουμε εδώ. Συμφωνούμε όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι να, προ, να προσπαθήσουμε για την μέγιστη δυνατή ε, συμβατότητα με αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, όσον αφορά τις εφαρμογές βασισμένα σε δορυφόρο, να τονίσουμε την, ε, τη σημασία αυτής της πτυχής, να τονίσουμε τη σημασία της έρευνας που έχει γίνει και να τονίσουμε την ανάγκη να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, ε, ιδιαίτερα στα στοιχεία για την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και σε αυτό το μέρος του προγράμματος και μάλλον να εστιάσουμε αποκλειστικά στις ε, πτυχές έρευνας και ανάπτυξης των εφαρμογών μεταφορών. Όμως, η αναγνώριση είναι ευρεία και πιστεύω ότι ο βαθμός σύγκλησης είναι πραγματικά μεγάλος. Επίσης, σημειώσαμε τα υπόλοιπα σχόλια και τις προτάσεις από εσάς που μόλις ε, μιλήσατε και πραγματικά ε, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρίσπεκ. Ε, κυρία Γκρίσπεκ, κάτι που θέλετε να προσθέσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους και για τα στοιχεία που συνείσφεραν και που θα τα εκπονήσουμε από κοινού. Και τους ευχαριστώ επίσης για τη συνολική υποστήριξή τους. Και σας ευχαριστώ επίσης για αυτή την ιδέα της υπεραξίας που θα μπορούσαμε να εκφράσουμε στον τομέα των μεταφορών μέσω αυτού του φακέλου μας, αυτής της έκθεσης. Σημείωσα δε όλα τα σχόλια που αναφέρεται όπως και τα παραδείγματα για την δυνατότητα εμβάθυνσης ε, της οργάνωσης των μεταφορών με τους νέους στη Γερμανία και αυτής της ιδέας, ε, της συνύπαρξης και να επικεντρωθούμε στα αστικά κέντρα. Επίσης, ε, αναφέρθηκαν και τρία πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία από την κυρία Ντιράν σε σχέση με το να δούμε και το θέμα ε, της ε, ζήτησης πέρα από τις προσφοράς ε, και επίσης αυτό το θέμα της υπεραξίας που αναφέρθηκε και από τον συναδελφό μου. Άκουσα τις παρατηρήσεις και τις κομισιόν, θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη, Πρόεδρε, καθώς ε, έχουμε κάπως καθυστερήσει χρονικά. Θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη προθεσμία για τις τροπολογίες για να έχω περισσότερο χρόνο να εργαστώ. Γιατί η παρουσίαση της ίδιας της έκθεσης αναβλήθηκε από τη μία συνεδρίαση στην άλλη της Επιτροπής μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να έχουμε μία προθεσμία για την κατάσταση τροπολογίας για τις 23 Αυγούστου. Έτσι θα είχαμε περισσότερο χρόνο για να εργαστούμε ακόμη περισσότερο και να έχουμε μια πιο ποιοτική έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρίσμπεκ, ε, έχω σημειώσει ε, λοιπόν ότι η προθεσμία θα είναι 23 Αυγούστου για την κατάσταση τροπολογιών. Αν είναι κανείς εδώ τον Αύγουστο, τέλος πάντων αυτή είναι η προθεσμία που ορίζουμε και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 17 Σεπτεμβρίου και 18 θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή και κατόπιν στην Ήτρε θα έχουμε την ψηφοφορία τον Οκτώβριο. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε πιο αργά από αυτή την ημερομηνία και θα έχουμε συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Νοέμβριο. 23 Αυγούστου λοιπόν για τις ε, προθεσμ... η προθεσμία για τις τροπολογίες, με συγχωρείτε. Εντάξει, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Πρόκειται για τη μελέτη σχετικά με την ε, ασφάλεια των εναέριων εμπορευματικών μεταφορών. Ο κύριος Μακάριο είναι εδώ. Η κυρία. Η κυρία. Uh, uh, Η μελέτη αφορά την ασφάλεια ενέργειων πραγματικών μεταφορών από τις τρίτες χώρες. Ζητήθηκε τον περισμένο Ιούλιο από την Επιτροπή και υλοποιείται από ε, μια πορτογαλική Ένωση και έχουμε την ε, κυρία Μακάριο, η οποία είναι καθηγήτρια από την MPT. Αν ε, μπορείτε παρακαλώ να πάρετε το λόγο για 15 λεπτά, σίγουρα θα με βοηθούσε γιατί θα έχουμε και ρωτήσει από τους βουλευτές. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω εδώ τη μελέτη αυτή. Η μελέτη συνίσταται σε μια ανάλυση των ε, θεμάτων ε, της ασφάλειας των ε, ενέργειων εμπορευματικών μεταφορών από τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν, ο λόγος για την υλοποίηση αυτής της μελέτης έγκυται σε τρία τινά. Καταρχήν, στο ότι η ε, εναέριες εμπορευματικέ μεταφορές γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικές ε, στο πλαίσιο των εναερίων μεταφορών αλλά και ε, λόγω της, της τροπικής, διατροπικής εκτανομής που γίνεται στον τομέα των εμπορευμάτων και οι εναέριες μεταφορές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη παρουσία και στο θέμα ε, των ε, εμπορευμάτων, εμπορευματικών, μάλλον και στο πλαίσιο των εμπορευματικών ε, πτήσεων αλλά και των επιβατικών πτήσεων. Υπήρχε λοιπόν ε, μια μεγαλύτερη ανησυχία σε ό,τι αφορά των επιβατών. Έτσι λοιπόν επικεντρωθήκαμε και στους επιβάτες και ο τελευταίος λόγος ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις που ε, είχαν ε, θέσει ως στόχο κάποιες εμπορευματικέ μεταφορές και έτσι λοιπόν ε, χρειάστηκε να γίνει κάποια ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζεται να γίνει κάποια ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα έχει τρεις στόχους η μελέτη που μας ζητήθηκε. Καταρχήν να γίνει η αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εμπνευματικών μεταφορών. Ο δεύτερος στόχος ήταν να γίνει μια αξιολόγηση των μέτρων που προτείνονται για την ενίσχυση της ασφάλειας στις εμπνευματικές μεταφορές και τέλος να εντοπιστούν οι ευκαιρίες οι δυνατότητες για να διορθωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και η εφαρμογή του έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική βελτίωση ε, στην ασφάλεια των εμπερευματικών μεταφορών εναερίως. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε έγκυτο στου εξή τομεί. Καταρχήν έγινε μια πρώτη αναθεώρηση εις βάθος όλης της νομοθεσίας ε, σχετικά με τις ενέργειε μεταφορέ και συγκεκριμένα με τις μεταφορέ των εμπερευμάτων. Επίσης μια βιβλιογραφική αναθεώρηση επιστημονικού χαρακτήρα σχετικά με θέματα ασφάλειας και με θέματα κινήτρων αλλά και συμπεριφορές οικονομικών φορέων και από εμπειρική σκοπιά ε, προστρέξαμε σε τρεις πηγές ε, πληροφοριών. Ε, ένα σύνολο συνεντεύξεων και εμπειρογνωμόνων του τομέα, τους απευθυνθήκαμε στους stakeholders, ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε στα κράτη-μέλη και απαντήθηκε από μια μεγάλη ομάδα κρατών μελών και ένα σύνολο case studies που παρουσιάζουν τις διάφορες πραγματικότητες ε, που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν με αυτά καταλήξαμε σε δύο πορίσματα. Αφενός ε, το ποιο είναι η κατάσταση των σημερινών πρακτικών ε, και δεύτερον ποια είναι οι πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται και με ποια όση επιτυχία. Έτσι λοιπόν από την ρυθμιστική σκοπιά έχουμε διάφορες οντότητες που ασκούν μια επιρροή από νομοθετική σκοπιά. Πρώτη οντότητα είναι φυσικά η Διεθνής ε, Οργάνωση ε, της ε, Αεροπλοείας, ο ΙΚΑΟ. Ο ρόλος του ΙΚΑΟ ήταν να συστήσει ένα σύνολο γενικών κανόνων για να εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί από τα κράτη-μέλη. Αν το μεταξύ όμως, η ίδια η ε, διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία απόφασης ε, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει καθολική συμφωνία μεταξύ των διαφορών χωρών. Είναι αργή λοιπόν αυτή η διαδικασία και δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και πολλές φορές ε, χάνεται η ευκαιρία εφαρμογής καθώς καθυστερούν οι διαδικασίες. Στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ επίσης υπάρχει και ένα πρόγραμμα ελέγχου που επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ε, της ε, εφαρμογής, της συμμόρφωσης, αλλά δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά την εξαναγκασμό της συμμόρφωσης ή να εξασφαλίσει μία εφαρμογή καθώς έχουμε σύσταση και όχι ε, νομοθεσία υποχρεωτικού χαρακτήρα. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύνολο βασικών κανόνων που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συναπόφασης και κατόπιν έχουμε ε, εφαρμοστική νομοθεσία που υιοθετήθηκε μέσω της επιτροπολογίας και κατόπιν Έχουμε και τα κράτη-μέλη που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και λαμβάνουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα ως προς την εφαρμογή στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών ε, βλέπουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Ευρώπη. Έχουμε μια υπηρεσία ασφάλειας, ένα οργανισμό ασφάλειας για τις μεταφορές, τη TSA, και ε, ο οργανισμός αυτός εκδίδει συγκεκριμένους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλες τις πτήσεις ε, με προορισμό αμερικανικά αεροδρόμια. Υπάρχουν και εγκαταστάσεις που εγκρίνονται από την TSA. Έτσι λοιπόν έχει δικαιοδοσία ο οργανισμός ε, για να αξιολογεί και να εγκρίνει τις εγκαταστάσεις και η ρύθμισή της ε, καλύπτει, μάλλον επεκτείνεται και πέρα από την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, ε, σε βιομηχανικό επίπεδο, σε επίπεδο του κλάδου, έχουμε την αυτορύθμιση. Έχουμε ε, την περίπτωση της ΕΑΤΕΜ που έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας και κυρίως στο επίπεδο των επισήμων ελέγχων. Και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τις μεταφορές επιμελητίας. Ε, έχει ήδη εκπονήσει ένα ε, χειρίδιο συστάσεων ε, για τις ε, αλυσίδες εφοδιασμού. Και θα ήθελα να τονίσω, και συγγνώμη που το λέω μόνο τώρα, ότι όταν μιλώ για ε, ασφάλεια αναφερόμαι στο security και όχι στο safety, γιατί έχουμε μόνο μία λέξη στα πορτογαλικά. Λοιπόν, πώς ε, έχουν τώρα οι διαδικασίες ε, ασφάλειας ενέργειων εμπορευματικών μεταφορών στον ευρωπαϊκό τομέα ουσιαστικά. Έχουμε δύο είδη διαδικασιών. Ε, καταρχήν έχουμε ασφάλεια της λυσίδας εφοδιασμού αλλά έχουμε και τη δειγματοληψία των εμπορευμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία της ασφάλειας της λυσίδας ευδιασμού, οι έλεγχοι γίνονται από τη στιγμή που τα έχουν κλείσει, δηλαδή από τη στιγμή που έχει κλείσει η αποστολή και γίνεται καθόλου το μήκος της αλυσίδα και βασίζεται στο διαδικασία της πιστοποίησης όλων όσων συμμετέχουν ε, σε αυτή την αλυσίδια του εφοδιασμού. Τώρα έχουμε και τη διαδικασία της δειγματοληψίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που συνήθως ε, γίνεται στο ίδιο το αεροδρόμιο στο χώρο του αεροδρομίου, δηλαδή δεν καλύπτει όλη την λυσίδα εφοδιασμού και πρόκειται για μία μέθοδο που λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζεται ανάλογα με τη φύση του ίδιου του εμπορεύματο. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένε περιπτώσει, στην περίπτωση των ΗΠΑ ε, και στι πτήσει με προορισμό τη ΗΠΑ, είναι η μόνη μέθοδο που γίνεται αποδεκτή. Έχουμε αυτέ τι δύο λοιπόν μεθόδου, αν θέλετε, που υλοποιούνται παράλληλα και εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Κατόπιν έχουμε διαδικασίες που εφαρμόζονται για πτήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες ε, με προορισμό την Ευρώπη. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και ένας από τους στόχους αυτής της μελέτης είναι ακριβώς να αξιολογήσει αυτή τη ρύθμιση που πρόσφατα έχει τεθεί σε εφαρμογή και μάλιστα έχει τροπο, θα τροποποιηθεί από το 2014. Από το Φεβρουάριο του 2012 έχουμε ένα σύνολο φορέων, έχουμε ένα σύνολο εταιριών που θα Ε, που θα πρέπει να ε, παρουσιάσουν και να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν κάποια σχέδια ασφάλειας για τη μεταφορά εμπορευμάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν ε, μιλάμε για την πιστοποίηση ECC3 και από τον Ιούλιο 2014 έχουμε μία νέα τροποποίηση. Αυτά τα σχέδια ασφαλείας και διαδικασίες θα είναι αντικείμενο ανεξάρτητης αξιολόγησης. Δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2014 έχουμε ε, την ευθύνη ε, της εταιρεία και από τον Ιούλιο του 2014 και μετά θα έχουμε μια ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης για κάθε συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ειδική για κάθε αεροδρόμιο. Έτσι λοιπόν το να ε, διασφαλιστεί η συμμόρφωση ε, θα χρειαστεί για να γίνει αυτό κάποια εκχώρηση σε ορισμένε χώρε, ενώ σε κάποιε άλλες χώρε ε, θα υπάρξουν πιο αυστηρές διαδικασίες Έτσι λοιπόν θα υπάρξει και μία ανάλυση κινδύνου που θα σχετίζεται με το με ποια χώρα πρόκειται αλλά και θα υπάρχουν και, και άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα ποιες είναι οι κυρίες ανησυχίε που μπορέσαμε να εντοπίσουμε σε αυτή τη μελέτη. Είτε ακούγοντας ε, τους ε, διάφορους ε, φορείς, είτε εξετάζοντας τις ίδιες διαδικασίες. Βρήκαμε ένα παράδειγμα ασφάλειας, το οποίο έχει διατυπωθεί στις ε, μεταφορές, έχει σχηματιστεί μάλλον στις μεταφορές των επιβατών και προσανατολίζεται για την αξιολόγηση του κινδύνου από εξωτερικές απειλές. Όλο αυτό το παράδειγμα ασφάλειας λοιπόν έχει ε, υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές απειλές. Έχουμε κάποια πρότυπα και κάποιες ρυθμίσεις έχει αυξηθεί η διοικητική πολυπλοκότητα και αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί και το κόστος υλοποίησης των δράσεων. Και φυσικά κατόπιν ε, πρέπει να καλύπτονται από τις διάφορες εταιρείες ε, αυτές οι πρόσθετες δαπάνες. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε και την ικανότητα των διαφόρων αρχών στα διάφορα κράτη-μέλη. Βρήκαμε σημαντικές αποκλήσεις σε ό,τι αφορά ε, το πόσο τα διάφορα κράτη-μέλη γνωρίζουν τις ίδιες διαδικασίες. Και επίσης βρήκαμε αλλαγές σε σχέση με τα αποκαλούμενα προγράμματα του ε, γνωστού αποστολέα και αυτό ουσιαστικά βελτίωσε την ανταλλαγή ε, πληροφοριών ε, σε όλη την αλυσίδα. Όμως ε, τελικά τι είδαμε, ότι τελικά υπήρξε μείωση αυτής της συνεργασίας γιατί κάθε φορά υποστηρίζονταν από τεχνολογικές λύσεις σε σχέση με μία μέθοδο για την ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πτήσεις ε, εισόδου, είδαμε και εκεί μία σειρά ανησυχιών που κυρίως έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας σε ορισμένες χώρες και σε πολλές περιπτώσεις είδαμε να μην εφαρμόζονται παρκώς οι κανόνες του ΙΚΑΟ, δηλαδή το επίπεδο της ε, εφαρμογής και η ίδια η στάση της κάθε χώρας ε, σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων του ΙΚΑΟ ε, ήταν διαφοροποιημένη. Υπάρχει λοιπόν κάποια έλλειψη εναρμόνισης εδώ και επίσης διαπιστώσαμε ότι ο ΙΚΑΟ λόγω της ίδιας της φύσης του δεν είχε την ικανότητα να μπορέσει να αντιδράσει γρήγορα έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι. Επίσης, οι αεροπορικές εταιρείες είχαν δυσκολία στο να διασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και στην πραγματικότητα, στη νέα νομοθεσία δεν βρήκαμε μία ανάλυση κόστους ωφέλους που να μας επιτρέπει να έχουμε μία πιο συγκεκριμένη ανάλυση του αντικτύπου σε ό,τι αφορά το κόστος ή να δούμε ποιο θα είναι το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα ή ποιο θα είναι το κόστος του να μην έχουμε τροποποιήσεις. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα νέο στρατηγικό όραμα για την ομοθεσία ε, που θα διέπει την ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ή διαδικασίες ασφαλείας θα πρέπει να προσανατολιστούν προς μια αξιολόγηση κινδύνου και όχι προς μια διοικητική διαδικασία. ή κανόνες θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη μεταξύ ε, της αξιολόγησης των εσωτερικών και των εσωτερικών απειλών και θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις ανησυχίες και τις διαδικασίες ε, από την πλευρά των επιβατών και θα πρέπει να δημιουργηθούν και κάποια κίνητρα για την έρευνα και για τις επενδύσεις στα συστήματα ασφαλείας και στους εξοπλισμούς. Στην αναβάθμιση λοιπόν των εξοπλισμών. Επίσης πρέπει να προωθηθεί μια συνεργασία μεταξύ ε, των επιχειρηματικών εταίρων και να διασφαλιστεί ότι ο ρόλος των αρχών ενισχύεται σε επίπεδο εποπτείας της ασφάλειας. Ουσιαστικά δηλαδή τι, ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε εδώ με αυτή την αλλαγή προσανατολισμού ή με αυτή την αλλαγή παραδείγματος ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εναέριων εμπορευματικών μεταφορών. Είναι αυτό που μας δείχνει αυτό το διάγραμμα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι αυτή που βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα με πράσινο, δηλαδή έχουμε μια διάδοση των προτύπων, έχουμε αποτελεσματικότητα σχετικά μειωμένη έναντι των κόστους και των ε, επενδύσεων που πρέπει να γίνουν να διατηρήσουμε τις διαδικασίες αυτές και έχουμε μία απόπειρα μεταφοράς των ευθυνών. Δηλαδή, οι σημερινές διαδικασίες διασφαλίζουν ότι η ευθύνη μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο. Δεν διασφαλίζουν ότι υπάρχει μία συνολική ευθύνη μεταξύ των διαφόρων φορέων. Αν όμως δεν κάνουμε τίποτα, διατηρούμε την ε, μακροπρόθεσμη διαδρομή που βλέπουμε βλέπετε ε, με το ροζ χρώμα, δηλαδή θα διατηρήσουμε μία ε, ευθύνη περιορισμένη, θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή τη διαδικασία του push and pull της ανάληψης ευθύνης ε, μεταξύ των διάφορων αρμοδίων φορέων και μια εναρμόνιση των κανόνων. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση ε, όπου θα έχουμε τη διασφάλιση της ασφάλειας με ένα γραφειοκρατικό ε, χαρακτήρα, αλλά θα υπάρξει διάδοση των διάφορων προτύπων και αυτό θα σημαίνει υψηλό κόστος των διαδικασιών ασφαλείας. Τι ε, πιστεύουμε εμείς ότι είναι πιο χρήσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο αποτελεσματικό. Είναι να κάνουμε την αλλαγή για όσα βλέπετε στα πράσινα κουτάκια και να έχουμε μια ασφάλεια που θα προσανατολίσετε λιγότερο σε ένα συμβατικό ορισμό και θα περάσουμε στο να έχουμε διαδικασίες πιο συνεργατικές μεταξύ ε, των διάφορων ε, φορέων και επιχειρήσεων και θα έχουμε ε, η τυποποίηση και τη γνώση που θα περνά από την αλυσίδα της ασφάλειας και θα ξεκινάμε στην αποδέση ευθυνών από την επιλογή του προσωπικού. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει καλύτερη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων φορέων και είναι απαραίτητο να έχουμε ορισμένες διαφορετικές αλλαγές που να μπορούν τελικά να καλύψουν τα ζητήματα αυτά και να μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο. Ποιες είναι οι δράσεις, το κείμενο που παρουσιάσαμε παρουσιάζει κάποια πολιτικά μέτρα, θα παρουσιάσω εδώ ορισμένε από τις δράσεις που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες και είναι δυνατές να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσεγγίσει αυτές τι συγκεκριμένε ανησυχίες στην εφαρμοστική έκθεση της Οδηγίας 300-2008, περιλαμβάνοντας τη σημερινή κατάσταση εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ των διάφορων χωρών και μεταξύ των διάφορων ε, ε, εμπορευομένων και να αναλύθουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς μία διαδικασία ε, που θα είναι πιο συνεργατική και να αξιολογήσουν τις διάφορες διαδικασίες που εφαρμόζονται τους επιβάτες ε, προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των επιβατών και της ασφάλειας των εμπορευματικών μεταφορών. Ταυτόχρονα να ζητηθεί η αξιολόγηση αντικτύπου του νέου κανονισμού και επίσης ε, να αξιολογηθεί και το κόστος όχι μόνο της νέας νομοθεσίας αλλά και του να μην γίνει τίποτα και να υπάρξει και μια, ένας προσανατολισμός προς την ανάπτυξη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την έκθεση. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ περίπλοκο, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, έχει μεγάλη σχέση και με αυτό που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε από αυτά που μπόρεσα να διαβάσω από την μελέτη βλέπω ότι και στο μέλλον μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο ε, θα ασχοληθούμε με το θέμα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα και ίσως ε, έχουν σημειωθεί παραβάσεις και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Έπειτα, παρότι είναι μια ευρωπαϊκή πρόταση, ε, δεν θα έπρεπε να είμαστε μόνοι μας ε, με αυτή στον κόσμο. Η εκτίμηση, πιστε, εκτιμώ πως είναι... Εκτιμώ πως δεν πρέπει να είναι μόνο διοικητικό το ζήτημα, αλλά για μένα το ζήτημα της ευθύνης πρέπει να, και της αρμοδιότητας πρέπει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. για παράδειγμα η ευθύνη και θα μιλήσω με παράδειγμα το Βέλγιο, εάν η ευθύνη πηγαίνει από τον ένα στον άλλο και τότε πιστεύω ότι η διοικητική ασφάλεια θα έχει ελλείψεις. και το, το να σπρώχνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο δεν είναι η σωστή διαδικασία. Η αλυσίδα έτσι, δεν, ε, θα, η αλυσίδα έτσι θα σπάσει και πιστεύω ότι πραγματικά έχει έρθει η ώρα για να αναλυθούν ευθύνες, αλλά στην τελευταία, η τελευταία φάση της ε, μεταφοράς είναι πιστεύω αρκετά σημαντική, διότι ε, σε αυτό το τελευταίο στάδιο μπορούν, ε, μπορούν να πάνε πολλά πράγματα στραβά. Επίσης, να ε, ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει πιθανότητα αναγνω... Ε, η δυνατότητα αναγνώρισης. Να υπάρχει μια λύση για το σκάνινγκ των προϊόντων από κοινό επίπεδο, από κοινοτικό επίπεδο, διότι όταν η κάθε μία χώρα έχει διαφορετικές πρακτικές αυτό δεν βοηθά και πιστεύω ότι ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας η αναγνώριση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των ελέγχων. Αυτό για μένα είναι βασικό. Ελπίζω όμως ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και σε αυτόν τον τομέα, όπως ήδη αναφέρεται. Ε, ελπίζω να πάμε ένα βήμα παραπέρα και ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεγκράντα, ο εισηγητής μας. Μπορεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τόσο λεπτομερή ε, έκθεση που έκαναν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, όχι μόνο για τις απειλές, αλλά για την απογραφή της σημερινής νομοθεσίας και το πώς γίνονται οι έλεγχοι για τα φορτία στις εναέριες μεταφορές, αλλά και για τις προτάσεις. Θα ήθελα να καταθέσω μία σκέψη για να συμπληρώσω τα όσα είπε ο δικός μας εισηγητής και να σας πω πως στη δική μου έκθεση για την αεροπορική ασφάλεια μίλησα για τα μέτρα ασφαλείας για τους επιβάτες. Όμως, ξέρετε τι έγινε με το αεροπλάνο από την Ιεμένη το Δεκέμβριο του 2010. Και τότε σας ζήτησα στη δική μου την έκθεση να εντάξουμε και μέτρα για την ασφάλεια των εμπορευμάτων. Και έτσι ήταν πιο πλήρης η έκθεση από αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί αρχικά. Έτσι έγινε και κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεται σε αυτή την έκθεση είχαν ήδη συμπληρωθεί στην προηγούμενη έκθεση, δηλαδή ανάλυση κινδύνου για το πώς μπορεί να ελέγχεται το ταχυδρομείο και το φορτίο που θα πρέπει να είναι αναλογικό με την απειλή που παρουσιάζει η μεταφορά τους όταν το 38% ε, το αυτών μεταφέρεται σε ε, αεροπλάνα που επίσης μεταφέρουν επιβάτες. Μεγαλύτερη λοιπόν εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Συμμερίζομαι την ανάγκη ε, να παρακολουθήσουμε και τις συστάσεις του ΙΚΑΟ. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία ανάλυση πιο συγκεκριμένη ε, και από, σύμφωνα με τα όσα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012 και να εξασφαλίσει πως οι κανόνες που θα ακολουθούμε θα μας εξασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την ε, μελέτη που μας παρουσιάσατε. Όπως υπόθηκε και πριν από τον κύριο Πασκουάλ, ε, το σημαντικό είναι η ασφάλεια των επιβατών και έχουμε πει ότι τα εμπορεύματα, ο έλεγχο των εμπορευμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι στα αυτά τα εμπορεύματα υπάρχουν ε, κάποια δέματα ε, μέσα στα οποία βρέθηκαν εκρηκτικά. Η ασφάλεια λοιπόν των επιβατών είναι η μία πλευρά του νομίσματος, υπάρχουν από την άλλη τα εμπορεύματα που πρέπει να διακινηθούν και, αυτό είναι ένα, και το πρόβλημα αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα και σήμερα. Και εν μέρη έχουμε κάποιους ε, αξιόπιστους και μη αξιόπιστους ε, διανομή που πρέπει να ελεγχθούν. Είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο έλεγχο, όπω είπα. Επιπλέον, η έρευνα και η ανάπτυξη είναι άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι πηγαίνει καλά πώς μπορούμε να ε, βελτιώσουμε το σύστημα του σκάνινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο, στα εμπορεύματα και ποιες άλλες μεθόδους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ε, πέραν από αυτές που χρησιμοποιούμε τώρα. Και όσον αφορά την εναρμόνιση και την τυποποίηση, φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω όμως πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, διότι δεν έχουμε και πάρα... πρώτον δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεύτερον, η συνεργασία με τα, πάρα... με τα τρίτα κράτη ε, ε, μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα. Ε, βέβαια δεν ήθελα η μελέτη σας να παρουσιάσει περισσότερα ερωτήματα, όμως είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Όπως και να έχει όμως, πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντάντ. Ευχαριστώ πολύ. Καταγράφω καταρχήν δύο παρατηρήσεις. Αυτό που είπατε και εσείς κυρία μου, τι θα μας κόστιζε το να σταυρώσουμε τα χέρια αξιολόγηση κινδύνου. Θα ήθελα για τους επιβάτες να είχαμε εγκρίνει κάτι αντίστοιχο. Γιατί πιστεύω ότι για τους ελέγχους και για το θέμα των υγορών και τα λοιπά, το θέμα το οποίο θα πάει στην Επιτροπολογία, φοβάμαι πως εκεί είμαστε πολύ επίμονοι για το ότι πρέπει να ελέγχουμε το 100% των υγορών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είναι τεράστιο το κόστος για ένα κίνδυνο ο οποίο δεν ξέρουμε είναι πραγματικός. Το ίδιο και για τις μεταφορές νομίζω πως για παράδειγμα για, το, για τη μεταφορά κάποιων εμπορευμάτων όπως τα κομμένα λουλούδια για παράδειγμα δεν υπάρχει λόγος να μεταφέρονται έτσι και έτσι θα μπορούσαμε να ε, μειώσουμε και το κόστος. Με συγχωρείτε εκεί δεν θα πρέπει να ελέγχουμε κίνδυνο, θα μπορούσαμε λοιπόν να μειώσουμε έτσι το κόστος. Δεν είναι θέμα κανονισμού, δεν είναι θέμα πιστοποίησης διοικητικής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν για συνεργασία μεταξύ ατόμων. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε την εκπαίδευση και τις ε, ε, εργασίας του επίγειου προσωπικού γιατί πολλές φορές είναι λιγότερο καταρτισμένοι, αυτοί που χάνουν πιο εύκολα τη ζωή τους, ε, οι πιο ευέλικτοι και αν είναι τόσο ευάλωτο το εργατικό δυναμικό που μας ε, ε, που απασχολούμε, τότε είναι προφανές ότι οι διαταγές πολλές φορές δεν θα καταλήξουν στο σωστό πρόσωπο. Ξέρετε, με το γνωστό αποστολέα για παράδειγμα, με ένα γραφή ε, ή με, μια, με, ένα χαρτί, με μια ε, απλή υπογραφή καταφέρουμε να περάσουμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αξιολόγηση κινδύνου όχι μόνο για τα εμπορεύματα και τους επιβάτες, μείωση του κόστους για τα εμπορεύματα και αύξηση της ασφάλειας εκπαιδεύοντας το ε, επίγειο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να συνεργάζονται στην αλυσίδα πληροφόρησης που είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε μια επαρκή ασφάλεια στα αεροδρόμια μας. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Φώστερ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και, τον, και την καθηγήτρια για την παρουσίασή της. Δυστυχώ δεν είχα χρόνο να διαβάσω όλο το έγγραφο. Και επίσης ήταν αρκετά περίπλοκο δύσκολο να διαβάσω τις διαφάνειες, δεν μπορούσα να τις δω από εδώ. Όμως εντάξει πήρα, κατάλαβα το νόημα του, των όσων είπατε και της εκτιμήσης αντικτύπου. Δεν νομίζω ότι άκουσα κάτι πάρα πολύ διαφορετικό στο τέλος της παρουσίασης από αυτά που ξέρουμε ήδη. Δέκα χρόνια πριν ήμουν εισηγήτρια για την εναρμόνιση των αεροδρομίων στην Ευρώπη μετά τα γεγονότα της 11 η Σεπτεμβρίου, φυσικά στον τομέα της ασφάλειας. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια απλή απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Δεν, υπάρχει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια συνταγή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πασπαρτού. Υπάρχουν διαφορετικές απειλές ανάλογα με το κράτος και το κάθε κράτος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τα κατάλληλα μέτρα ασφαλεία, που αυτό ενδεχομένω να διαφέρει από κράτο σε κράτο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με ποιο έχει δίκιο και ποιο όχι, αλλά με τι συνθήκε και με αυτό που πιστεύει το κάθε κράτο ότι είναι το καλύτερο. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανονισμοί που ισχύουν και πρέπει να συμμορφωθούν ε, με αυτού του κανόνες. Όσον αφορά τον ε, ΙΚΑΟ, είναι ένα συμβουλευτικό σώμα, δεν έχει νομικό δικαίωμα να επιβάλλει ε, κανονισμούς, όμως τα περισσότερα κράτη-μέλη πιστεύω ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να συμμορφωθούν με ό,τι ήδη έχει, ε, έχει ισχύσει. Τώρα, πιστεύω ότι πριν δούμε καινούριου κανονισμού, πρέπει να κοιτάξουμε ότι υπάρχουν καλές πληροφορίε από τα κράτη-μέλη πίσω από αυτό Και όσον αφορά τους, ε, την ασφάλεια των επιβατών και των εμπορευμάτων υπήρξαν διάφορες, ε, διάφορα περιστατικά. Δεν συμφωνώ με την ε, κυρία Ζιράν ότι όταν κάποιο δουλεύει στον τομέα τη ασφάλεια είναι απαραίτητα και κακοπληρωμένο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι απάντηση στα προβλήματα τη ασφάλεια. Πάμε πέρα από αυτό. Όταν μια εταιρεία απασχολεί εργαζομένου και του απασχολεί για μια συγκεκριμένη δουλειά και έχουν κάποια συλλογική σύμβαση, η εταιρεία αυτή φροντίζει οι υπαλλήλοι τη να είναι καλά εκπαιδευμένοι. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει η δουλειά τους. Γενικά πιστεύω ότι το προσωπικό στα αεροδρόμια κάνει καλή δουλειά, όμως είναι η ευθύνη του αεροδρομίου, των αερομεταφορέων και των άλλων σχετικών για να συμμορφωθούν με όλε αυτέ τι απαιτήσει ασφαλείας. Επίσης, ε, τα τα, τα background check είναι ακόμα σημαντικό για τους υπαλλήλου που δουλεύουν εκεί και αυτό πώς θα το συνδέσουμε με την προστασία δεδομένων. Επίσης πρέπει να υπάρχει αναγνώριση, γιατί για παράδειγμα όταν κάποιος θέλει να δουλέψει σε, μια, σε έναν ευαίσθητο τομέα, οι προσωπικά δεδομένα θα ζητηθούν φυσικά, ίσως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους εργοδότες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι γενικά ένα δύσκολο και περίπλοκο θέμα για κάποια κράτη-μέλη. Ε, σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι οι λύσει που βασίζονται στην τεχνολογία είναι καλέ και πω προχωρούν συνέχεια. Δεν μπορούμε να, να βάλουμε όμω το φορτίο, ολόκληρο το φορτίο σε ανιχνευτή, κατά ανιχνευτή μετάλλων. Όμω, ε, ε, αναφερθήκατε στους, στους non-consigners και συζητήσαμε και για τις δημόσιες προμήθειες και για το πώς ε, μετακινούνται τα αγαθά και φυσικά ναι, είναι ένα θέμα το ποιος ξέρει ποιον, από πού έρχεται το κάθε τι, τι γίνεται. Μπορεί να έχουμε όντως κάποια ζητήματα με τρίτες χώρες. Όμως πολλές φορές ξέρουμε ότι φορτία έρχονται και πηγαίνουν σε χώρες οι οποίες έχουν πολιτική αστάθεια. Σε γενικέ γραμμέ, όμω, πιστεύω ότι ο καθένα κάνει το, το καλύτερο δυνατό για, για να υπάρχει ασφάλεια. Οι περισσότεροι μεταφορεί, αερομεταφορείς εμπορευμάτων κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Υπάρχει βελτίωση και γενικά πιστεύω ότι είναι καλό να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να δούμε τι ε, σχόλια θα έχει να κάνει η Κομισιόν στην εκτίμηση αντικτύπου της. Μια εκτίμηση η οποία είναι εκτενέστατη και πώς θα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Μάλιστα, η Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Αστρό Σνάιντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Εδώ συζητούμε για τις, ε, για τα, τις εμπορικές μεταφορές ε, με αεροπλάνο. Αυτό ας παραμείνουμε εκεί και ας μην αναφερθούμε στην ε, ασφάλεια. Δεν θα αναφερθώ τουλάχιστον εγώ στην ασφάλεια. Πιστεύω ότι από αυτά που μάθαμε μέσα από όλες αυτές τις συζητήσει για τους ε, ανιχνευτές για τα σκάνερ, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αρκετά καλό σύστημα όσον αφορά την αεροπορική ασφάλεια. Αντίθετα από άλλου τομεί, η βιομηχανία του τομέα αυτού βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση όσον αφορά ε, τα, τις, ε, τους μεταφορείς ε, των εμπορευμάτων, τα αεροδρόμια και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει περίπου 40 επιθεωρήσεις αεροδρομίων σε κράτη-μέλη, ασκεί ελέγχου ποιότητα, έχει τέτοια προγράμματα και φυσικά και αξιολογούμε την ασφάλεια και η εναρμόνιση έχει επιτευχθεί με τρόπο πραγματικά θαυμαστό τα τελευταία χρόνια στα αεροδρόμια. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε άρθρο 15 με το οποίο λέμε στα κρατημέλη του αεροδρομίου σας δεν είναι κατάλληλο να ε, μεταφέρει εμπορεύματα ή επιβάτες ε, προς το παρόν. Δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές. Η έκθεση αυτή λοιπόν, ναι, ίσως θα μπορούσε να τροποποιηθεί ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν τις, ε, τα κατάλληλα σχόλια ε, στους ε, επιμέρους τομείς που τους αφορούν. Κάποια στοιχεία μας τα παρουσιάσατε πολύ χειρότερα από, όσο τα έχουμε δει εμείς στις αποθεωρήσεις μας. Τώρα η ασφάλεια φυσικά ένα σημαντικό εργαλείο για την ασφάλεια που έχει εξάγει ο ΙΚΑΟ σε άλλες χώρες. σε πολλές τρίτες χώρες ε, χρησιμοποίησαν με χαρά τους αυτό το όργανο που δημιουργήσαμε και αναπτύξαμε εμείς και η, ε, η όλη βιομηχανία αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών ε, είναι πολύ πρόθυμη να κάνει αυτό το screening, αυτή την εξέταση του φορτίου στα αεροδρόμια. Και αυτή η εξέταση, αυτό το screening είναι, κάτι από τις, από τους, είναι ένας από τους πιο κρυβούς και δαπανηρούς ε, τρόπους ελέγχου. Επίσης, αναφέρατε ότι πρέπει να υπάρχει ε, περισσότερη ε, εκτίμηση κινδύνου. Υπάρχει νομοθεσία που εισήχθη τον Φεβρουάριο αυτόν τον καιρό, η οποία ήταν η εκτενέστατη που έχει γίνει ποτέ. Τα κράτη-μέλη βοήθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πληρέστατη εκτίμηση κινδύνου μαζί με τους συναδέλφους από την, τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, τους υπουργούς εσωτερικών και αυτή λοιπόν η πλήρη εκτίμηση κινδύνου έχει διεξαρθεί όσον αφορά την ε, αεροπορική εμπορευματική ασφάλεια και είναι, αποτελεί βάση για νομοθεσία. Εμεί συνεχίζουμε να τροποποιούμε και να προσαρμόζουμε με την νομοθεσία, να ε, κάνουμε εξαιρέσεις, να ε, εισαγάγουμε πιο αυστηρά μέτρα σχετικά με τη μεταφορά φορτίων με αεροπλάνο και πάντα βασιζόμαστε στις ε, πιο επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με, τις, τα προβλήματα ή με τα βάλωτα σημεία των αεροδρομίων στις τρίτες χώρες. Τέλος, εάν δεν είχαμε ένα τόσο εναρμονισμένο και συμπαγές σύστημα αυτό που έγινε ε, στην πρώτη... Ε, δεν θα είχε γίνει αυτό που συνεβεί στην 1η Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε συμφώνησαν με μηδέα αναγνώριση του καθεστώτος ε, μεταφοράς φορτίου με αεροπορικής μεταφοράς φορτίου να μεταφέρουν όλους τους διπλούς ελέγχους στα, ευρωπαϊκά, στα ενωσιακά αεροδρόμια από, σε φορτίο που πηγαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε, θα μεταφέρουν στα ε, ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Δεν θα είχαμε μια τέτοια συμφωνία αν το σύστημά μα δεν ήταν συμπαγέ και, και πλήρω αναμονισμένο και αν ο εταίρο μα δεν ήταν πεπισμένο ότι οι κανόνε μα εφαρμόζονται και είναι αποδοτικοί σε όλο τον ε, χώρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Μακάριο, θα ήθελατε να απαντήσετε στα σχόλια. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια αυτά. Εν γέννη συμφωνώ και αντικατοπτρίζονται ευρέως ε, στην έκθεση. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύπλοκης διαδικασία Ας είμαστε σαφείς. Προφανώς ε, η έννοια της ασφάλειας ε, της αλυσίδας εφοδιασμού είναι μια έννοια ενδιαφέρουσα, με ιδιαίτερη αξία όμως αυτή τη στιγμή το να τεθεί σε λειτουργία, το πώς τίθεται σε λειτουργία ε, είναι με λυπή τρόπο και δεν υπάρχει πλήρη συνεργασία από τους εμπνευμένους. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια αλλαγή παραδείγματος που θα περάσει από το να έχουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ όσων κάνουμε σίγουρα στις, σήμερα στις διαδικασίες για τους επιβάτες και στις διαδικασίες για τα εμπορεύματα. Γιατί ένα πολύ σημαντικό τμήμα των εμπορευμάτων αυτών μεταφέρονται σε επιβατικά αεροπλάνα. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτών των διαδικασιών. Από την άλλη, ε, επειδή ε, για να είναι μάλλον η έννοια της ασφάλειας ε, όχι μόνο ε, κάτι θεωρητικό αλλά να έχει και μία πλήρη εφαρμογή είναι απαραίτητο τα θέματα της ασφάλειας της ερμηνείας του κινδύνου της γνώσης του επιμερισμού του επίπεδου αρμοδιότητας να πηγαίνουν όσο το δυνατόν προς το πάνω μέρος ανάντι ε, της ε, αλυσίδας εφοδιασμού και να μην ζημιώνονται από διαδικασίες όπως ε, συμβαίνει παραδείγματος χάρη στη διαδικασία του account consigner και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω παρά μία ανάθεση της ευθύνης και μία μεταβίβαση της ευθύνης ε, με ε, μία αποτελεσματικότητα σχετικά μειωμένη σε ό,τι αφορά την πραγματική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολύπλοκου συστήματος, πρέπει να το προσεγγίσουμε ως εξή. Πρέπει να υπάρχει αλλαγή παραδείγματος και προσαρμογή του παραδείγματος στα σημερινά επιχειρηματικά μοντέλα και στις σημερινές επιχειρηματικές ανάγκες. Αυτό περνά από την εναρμόνιση τεχνολογικών απαιτήσεων ε, και ε, απαιτήσει ικανοτήτων των ανθρώπων που συμμετέχουν στο στα διάφορα στάδια των διαδικασιών και στις διάφορες διαδικασίες. Και επίσης πρέπει να κατανοούμε τον κίνδυνο με ένα αρμονισμένο τρόπο, να έχουμε αρμονισμένες μεθοδολογίες και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης όπου πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα ανεξάρτητα με το αν μας εξυπηρέτησε ε, ορθά ως τώρα και πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα μας εξυπηρετεί ως δυνατόν καλύτερα και ότι δεν θα αποτελεί άχθος ε, για τους εμπορευμένους, για τους οικονομικούς φορείς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ικανοί να μειώσουμε το κόστος, να αυξήσουμε ε, τον επιμερισμό των ευθυνών και μειώνοντας ε, είτε το άμεσο κόστος είτε το αμέσο κόστος. Να ευχαριστήσω λοιπόν την καθηγήτρια Μακάρη, κυρία Μακάριο, για τον τρόπο που παρουσίασε την έκθεσή της, αλλά και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, 20 λεπτά διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με την Task Force, την ομάδα δράσης για το τουρισμό. Λοιπόν, διακόπτουμε μέχρι τις 5.30 και μια και είστε όλοι εδώ να πω πως στις 6 Σεπτεμβρίου, 5η, 9 ώρα το πρωί μέχρι 6.30 το απόγευμα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Στις 5.30 λοιπόν.